liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Στο σημείο 1 έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις αλλαγής για το σημείο 12 και για το σημείο 13 συγκεκριμένα. λίγο ησυχία όμω, τώρα νομίζω ότι με ακούτε καλύτερα. Λοιπόν, στο σημείο 1, έγκριση της ημερήσια διάταξης, έχουμε κάποιες αλλαγές στο σημείο 12 και 13 της ημερήσια διάταξης. Αύριο στην ψηφοφορία θα πρέπει αυτά να ψηφίσουμε πρώτα. Εντάξει, αν δεν διαφωνεί κανείς, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη με αυτή την τροποποίηση που έγινε. Έχουμε τη συνήθι, το συνήθες ε, καθεστώς διερμηνίας, τις γλώσσες που ο συνήθως έχουμε στην Επιτροπή μας. Δεν έχουμε εστονικά και μαλτέζικα. Έχουμε όμως κροατικά. Την ε, επόμενη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου, θα κάνουμε μία επιπλέον συνάντηση, μία νέα συνάντηση της Επιτροπής μας για το θέμα της ε, εμπορίας εκπομπών συζητείται αυτή η πρόταση της Επιτροπής και θα είναι παρούσα και η Επίτροπος και οι εμπειρογνώμονες και θα έχουμε αρκετό χρόνο από τις 3 μέχρι τις 6.30 την επόμενη Δευτέρα στις 12 για να συζητήσουμε αυτή την πρόταση της Επιτροπής για τις εκπομπές, για την εμπορία εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος. Και την Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα, 13 Νοεμβρίου, θα έχουμε μια ακρόαση για τους ε, υποψηφίους, ε, για τον, τους διαδόχους του Τζον Ντάνι, από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης. Και μια τρίτη ανακοίνωση για το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ένα workshop στις 15 Νοεμβρίου από τις 9.30 το πρωί στην αίθουσα ASP 5Ε2 ε και στις 26 ε, Νοεμβρίου στην αίθουσα ASP 5Ε3 ε θα έχουμε άλλο ένα workshop για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Στη συνέχεια, στο σημείο 3, έχουμε την έγκριση των πρακτικών από τις συνεδριάσεις της 6 Σεπτεμβρίου και της 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4 για την εκλογή τρίτου αντιπροέδρου. Και εδώ θα ήθελα να δώσω λόγο στον Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, στις ε, εκλογές ε, μετά το πέρας της μισής θητείας του Κοινοβουλίου, όταν έλαβε ο Πρόεδρος τα καθήκοντά του, ε, είχαμε πει ότι θα έπρεπε να αλλάξει ε, ε, κάποια θέση αντιπροέδρου και να δώσουμε την δυνατότητα και σε μία συνάδελφο, μία γυναίκα συνάδελφο να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα. Ο Γιάννος Φούρδας έγινε, ανέλαβε καθήκοντα στην Τσεχία και επομένως υπάρχουν αλλαγές στις εθνικές αντιπροσωπείες και μπορώ τώρα να σας ανακοινώσω ότι έχουμε τη συνάδελφο Κρίστα Κλάς, ε, μια ιδιαίτερα ε, διακεκριμένη συνάδελφο που μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα. Πολλοί συνάδελφοι τη γνωρίζουν, ε, γνωρίζουν τις σημαντικές εκθέσεις που έχει συντάξει για τα βιοκτώνα και πολλά άλλα θέματα. Είναι πολλά χρόνια βουλευτή του Ευρωκοινοβουλίου και νομίζω ότι τώρα θα είναι πληρέστερο το Προεδρείο με μια τόσο ικανή συνάδελφο από το ΕΛΚ και ζητώ την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σας. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητά το λόγο. Θα έλεγα να δεχθούμε αυτή την πρόταση. Αφόσον υπάρχει μόνο μία πρόταση, μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοής. Να τη συγχαρούμε. Συγχαρητήρια στη συνάδελφο Κρίστα Κλάς. Ελάτε παρακαλώ κυρία Κλάς. Σας συγχαίρω. Σας συγχαίρω και εξ ονόματος ολόκληρης της Επιτροπής. Λοιπόν, χαίρομαι που είμαστε και πάλι πληρέστατοι στο Προεδρείο μας και μπορούμε να συνεχίσουμε τα καθηκοντά μας. Παρακαλώ, κύριε Κούκοβιτς. Είχατε ζητήσει το λόγο. Ε, ε, ε, Ζητώ συγγνώμη, πρόεδρε. Να σας ενημερώσω για κάτι ήθελα να δώσω μια πληροφορία στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Υπάρχει ένα περιστατικό καταστροφών στην Σλοβενία. Έχουμε πλημμύρες αυτή τη στιγμή ε, στην Σλοβενία. Έχουν ξεχυλίσει τα ποτάμια, έχουν βγει από την κήτη τους ε, και πολλά σπίτια, πολλές επιχειρήσεις έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, ε, ακόμη και οι κάτοικοι διατρέχουν κίνδυνο και ως μέλος της Επιτροπής ε, θεώρησα σκόπιμο να σας δώσω αυτή την πληροφορία. Είμαι πεπισμένη ότι θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό που πλήττεται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί συναδελφέ για την πληροφορία που μας δίνετε και βέβαια θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Και ελπίζω να μην υπάρξουν περαιτέρω καταστροφές. Ωραία, περνάμε στο σημείο, 4, στο σημείο 5 της σημερινής διάταξης, ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Εδώ ήδη έχουμε κάνει τη συζήτηση και ο εισηγητής είναι ο Ρίχαρτ Ζίμπε. Είχαμε καλέσει και εμπειρογνώμονες. Είναι παρούσα και η Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΙ και η Γενική Διεύθυνση, ΣΑΝΚΟ ε, δεν είναι αρμόδια και δεν ε, θέλει να παρέστη. Ε, και λόγω τεχνικών προβλημάτων ε, έχουν μείνει στην Αθήνα ε, στο αεροδρόμιο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο όμως στον εισηγητή, στον κύριο Ρίχαρτ Ζέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Κρίστα Κλάς και να πω ότι χαιρόμαστε που έχουμε και μια γυναίκα στο Προεδρείο γιατί πραγματικά είναι πληρέστερο το Προεδρείο. Θερμά συγχαρητήρια. Δεύτερον, θα ήθελα να εκφράσω την συμπάθειά μου και τη λύπη μου για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Σλοβενία και μας ανέφερε η συνάδελφος κυρία Κούκοβιτς ε, για τις πλημμύρες στη Σλοβενία. Έχουμε συζητήσει και την οδηγία για τις ε, πλημμύρες. Ήμουν και εγώ για την αποφυγή των φυσικών καταστροφών, και εγώ εισηγητής και ε, είναι ένα θέμα το οποίο συχνά μας απασχολεί. Λοιπόν, για την έκθεση αυτή, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, έχουμε κάνει ήδη μια συζήτηση. Έχουμε συζητήσει τα προθεσμία για τις τροπολογίες και ε, πολλοί συνάδελφοι υπέβαλαν τροπολογίες για την έκθεση αυτή Υπάρχουν πολλέ απόψει και προσπάθησα, λαμβάνοντα υπόψη τι τροπολογίε, να λάβω υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερε απόψει. Το συζήτησα και με του ε, εμπειρογνώμονε και ε, καλέσαμε και τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και εγώ και η κυρία Ροτ Μπέραντ, αλλά δεν μπόρεσε η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ε, να περαστεί. και η Προεδρία επίσης δεν μπορέσε να παραστεί γιατί λόγω των τεχνικών προβλημάτων έχουν μείνει στην Αθήνα. Θέλουμε να συζητήσουμε τα βασικά σημεία στα οποία ενδέχεται να υπάρχουν ε, κάποιες ε, διαφωνίες και να υπενθυμίσω ότι στο πλαίσιο, στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα η Επιτροπή μιλά για αυτόν τον κατάλογο των ε, ουσιών προτεραιότητας και για τη συμπλήρωση αυτού του καταλόγου. Αυτές ήταν οι προτάσεις της Επιτροπής και θα ήθελα να σας υπενθυμώσω ότι δεν πρόκειται καταρχήν για, τα, για το πόσιμο είδωρ και για την ανθρώπινη υγεία. Περισσότερο πρόκειται για τα επιφανειακά βασικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θέλουμε να διατηρήσουμε σε καλή ε, χημική κατάσταση μέχρι το 2015. Από τις 33 ουσίες, οι 15 πέρασαν από τις προτινόμενες 33 δηλαδή, ουσίες και η Επιτροπή ξεκίνησε μία μακρά επιστημονική διαδικασία. Στις διάφορες συζητήσεις παρέστησαν και εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη και από τους ενδιαφερομένους και προτείνεται τελικά αυτός ο κατάλογος ουσιών. Εδώ έχουμε μία πρόταση που είναι επαρκώς επιστημονικά βασισμένη. Ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες μελέτες σε αυτή την αξιολόγηση από ομοτύπους, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να βασιστούμε στα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα στην ε, που έχουμε μέχρι τώρα διαθέσιμα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Φαρμακευτικά προϊόντα, φαρμακευτικές ουσίες οι ουσίες φαρμακευτικής σημασίας μπαίνουν στα επιφανειακά ύδατα και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέτες ε, αυτό τεκμηριώνεται και πρέπει να δούμε εάν ε, ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις για το περιβάλλον όσον αφορά αυτές τις φαρμακευτικές ουσίες. και αν πληρούνται τα ε, πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος ε, τα οποία έχουν ε, τεθεί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος ε, μετατροπής της νομοθεσίας και το κόστος ε, μη μετατροπής ε, και να λάβουμε υπόψη μας και τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 191 της συνθήκης. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την μετατροπή και γι' αυτό υπάρχουν κάποιες πολιτικές αδυναμίες σε αυτή την πρόταση και θα πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα που εμπλέκουν και θέματα κόστους να συζητηθούν στο Συμβούλιο πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι ουσίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο και να δούμε κατά πόσο υπάρχει αναλογικότητα με το κόστος το οποίο συνεπάγονται αυτές οι διατάξεις. Υπάρχει μία σουηδική μελέτη που μιλά για το ε, κόστος που μιλάει για 17 έως 19 ευρώ ανά άτομο ανά έτος και υπάρχει και μια άλλη μελέτη ε, όπου δεν ε, αναφέρονται μόνο οι τρεις βασικές φαρμακευτικές ουσίες αλλά και περισσότερες φαρμακευτικές ουσίες ε, και γίνεται και πιο μακροπρόθεσμη ανάλυση των επιπτώσεων αυτών των χημικών ουσιών και τις επιπτώσεις για τη στιβάδα του όζοντος και πρέπει να δούμε πότε θα θεσπιστεί αυτό αυτή η οδηγία. Η δικλοφενάκη, παραδείγματο χάρη, είναι μια ουσία που μπορεί να παραμείνει στον κατάλογο, να αλλάξει η ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να πληρούνται τα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί. ώστε να φτάσουμε στα τελικά πρότυπα το 2026 το Συμβούλιο αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ότι υπάρχει πλειοψηφία των κρατών μελών κατά της πρότασης να μπουν στον κατάλογο αυτές οι ουσίες. Και νομίζω ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλές ε, αντιρρήσεις ε, κατά της πρότασης αυτής. Υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος, όπως είπαμε, υπάρχουν δεδομένα τα οποία πρέπει να πληρούνται. Δεν έχουμε τεράστιες αλλαγές στον κατάλογο. Υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ ενός δεσμευτικού καταλόγου. Μια ουσία πρέπει να παραμένει στον κατάλογο τέσσερα χρόνια κατά μέγιστο όριο και θα πρέπει να ελεγχθεί ε, η συγκέντρωση της ουσίας αυτής στα ύδατα μετά από τρία χρόνια. Πολλοί φοβούνται ότι θα είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος της επιτήρησης. Όσον αφορά ε, το θέμα της ασφάλειας ε, από πολιτικής πλευράς είναι ενδιαφέρον και το θέμα των cross-links, δηλαδή ε, υπάρχουν προϊόντα τα οποία νομίμως βρίσκονται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προϊόντα παρασιτοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, βιοκτόνα, υπάρχουν προϊόντα τα οποία ρυθμίζονται από άλλη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ πρέπει να δούμε ε, τη σχέση μεταξύ μιας επίσημης έγκρισής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, του προβλήματος που μπορεί να προκαλούν στα επιφανειακά ύδατα. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις σχετικές απόψει, γιατί όταν ε, μια ουσία φτάνει ένα, ξεπερνά ένα κατόφλι στα επιφανειακά ύδατα δεν σημαίνει αυτό αυτόματα ότι αποσύρεται η αδειοδότηση του προϊόντο. Είναι διάφορα θέματα λοιπόν που πρέπει να συζητηθούν αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ ε, των στοιχείων που πρέπει να ρυθμίσουμε. Υπάρχει η πολιτική για τα ύδατα και η πολιτική για την υγεία των κρατών μελών. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς εδώ με την πολιτική για τα ύδατα να ρυθμίσουμε θέματα που άπτονται της πολιτικής υγείας. Υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες σε κάποια σημεία. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να βρούμε ένα ισορροπημένο μείγμα διατάξεων. Αυτά λοιπόν και ευχαρίστω να συνεχίσουμε τη συζήτηση με όποιον συνάδελφο θέλει να κάνει ερωτήσει. Ευχαριστούμε κυρία Ζέβα. Δεν έχουμε κάποιο εκπρόσωπο από τη Σουηδία. Αναφέρθηκε όμω ήδη η μελέτη αυτή ε, από τη Σουηδία. Νομίζω ότι την έχετε την μελέτη ω παράρτημα στα έγγραφά σα και έχουμε ε, νομίζω και κάποιον εκπρόσωπο από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα μπορούσαμε ε, να θέσουμε τι ερωτήσει αυτέ. Πριν σας δώσω το λόγο, να δώσω το λόγο στην Επιτροπή Πέτερ Γκάμελτοφ, που είναι επικεφαλής της Μονάδας Προστασίας των Ιδάτινων Πόρων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία να σας εξηγήσω κάπως ποιο είναι το ιστορικό αυτής της πρότασης. Έχει γίνει μία συζήτηση και γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος όσον αφορά το γενικό ε, ιστορικό. Ο στόχος είναι η ανανέωση της οδηγίας 2008 κάθετος 105 που απαριθμεί τις ουσίες προτεραιότητας και ορίζει τα περιβαλλοντικά πρότυπα ε, για αυτές τις ουσίες. Έχουμε κάνει, έχουμε μελετήσει μεγάλα προγράμματα για να εντοπίσουμε τα προγράμματα τα οποία έχετε τώρα ενώπιον σα. Είχαμε 2.000 ουσίες στην αρχή, σιγά σιγά μειώθηκαν ε, μέσω διαδικασιών των ακαδημαϊκών συμμετεχόντων και των κρατών μελών. Έγιναν αξιολογήσεις από την Ενεξάρτητη Επιτροπή Επιστημονική Επιτροπή της ε, Κομισιόν όσον αφορά τις ε, ουσίες και οι 15 ουσίες επελέχθησαν διότι υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η συγκέντρωση αυτών των ουσιών ξεπερνά τα επίπεδα ασφάλειας. Η γνώμη μας είναι ότι δεν θα πρέπει αυτό να το θάψουμε κατά κάποιο τρόπο, να το αποσιωπήσουμε, αντιθέτως θα πρέπει να το μελετήσουμε και να το διερευνήσουμε. Από τη στιγμή που υπάρχει λόγος ανησυχίας για άλλες ουσίες, θα πρέπει να βελτιωθεί η βάση δεδομένων και η βάση γνώσεων όσον αφορά την διάδοση των ουσιών αυτών στο περιβάλλον και έπειτα υπάρχει και το θέμα των πανταχού παρουσών, όπως αποκαλούνται ουσίες, που δηλαδή Εξακολουθούν να υπάρχουν στο περιβάλλον διάφορες ουσίες και έχουμε κάνει προτάσεις ώστε να σημειωθεί πρόοδος παρά τις ουσίες που μας ενοχλούν και που υπάρχουν στο περιβάλλον μας για χρόνια και θα συνεχίσουν να υπάρχουν για χρόνια ακόμη. για το θέμα του κόστους και των φαρμακευτικών Αυτά είναι τα βασικά θέματα που συζητώνται εδώ. Καταρχήν, όπως είπε ο κύριος Σίμπερ, ε, καταρχήν υπάρχει θέμα υπά... σύνδεσης με τα βιοκτώνα, τα ζανιοκτώνα, την ε, νομοθεσία περί φαρμακευτικών προϊόντων και ούτω καθεξής. Ο βασικός κανόνας ε, είναι ότι τα κρατημέλη στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισής τους θα είναι αυτά που θα αποφασίσουν ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Οποιαδήποτε εκτίμηση γίνει από πλευρά της Κομισιόν ε, γίνεται με την εν ε, γνώση του ότι δεν ξέρουμε τελικά ποια κράτη ε, θα αφορούν αυτές οι πληροφορίες. Για τα φαρμακευτικά προϊόντα οι πληροφορίες είναι από την Ελβετία και κάποιες πληροφορίες είχαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε επίσης κάποιες πληροφορίες από τη Γερμανία για το κόστος της αφαίρεσης συγκεκριμένων ουσιών από τον χώρο ρήψης ε, αποβλήτων. Και τα στοιχεία επίσης που έχουμε είναι στι αξιολογήσεις που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη. Και άρα Επ' αυτών των πληροφοριών που μας δώσαν τα κρατημέλη έχουμε κάνει και εμείς τις αξιολογήσεις μας και από αυτά που είναι διαθέσιμα από το, την, ε, υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και τη Eurostat. Ξεκινήσαμε... Υπάρχει φυσικά λόγος για ανησυχία. Το κόστος που αναφέρεται εδώ είναι το maximum κόστος γιατί αναφέρεται στην ε, ε, επεξεργασία αποβλήτων, οι επιλογές και η πρόληψη φυσικά θα οδηγήσουν στη μείωση του κόστους. Πρόληψη μπορεί να είναι οι φράχτες, για παράδειγμα για, τον τη διαχείριση των ιστρογόνων, είναι οι φράχτες για τα ζώα, όπως γίνεται και με τις ορμόνες ας πούμε να υπογραμμίσω ότι η Κομισιόν δεν περιορίζει την υγειονομική περίθαλψη ή την χρήση αντισυλληπτικών. Αυτό όμως που προτείνουμε είναι να αναζητήσουμε την λιγότερο δαπανηρές λύσεις. Η πρόληψη θα περιορίσει δε τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται ειδική αγωγή ε, όμως τα προβλήματα αυτά προκύπτουν και λόγω των δημογραφικών αλλαγών ε, και λόγω των οικονομικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών, πολύ σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι ε, καθορίζουν το είδος της ε, αγωγής που χρειάζεται. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω αγωγή ή κατεργασία. Εφόσον ε, γίνει σωστά η πρόληψη θα περιοριστεί και το κόστος κατά συνέπεια. Να σας αναφέρω ότι έχουμε ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για το νερό με στόχο να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και στην παροχή λύσεων για αυτού του είδους περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μάλιστα, η κατεργασία λιμάτων ε, είναι ένα πρόβλημα και πολύ σοβαρό, πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Θα ε, ελπίζουμε πως αυτή η εταιρική σχέση καινοτομία θα μας δώσει λύσεις, ε, γιατί σαφώς βρισκόμαστε σε ένα τομέα όπου δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία και όπου σίγουρα οι τεχνολογικές εξελίξεις θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους. Τέλο, να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι η οδηγία πλαίσιο για το είδωρο δίνει στα κρατημέλη αρκετή ευελιξία, δίνει την ευελιξία να αναβάλουν, δίνει την ε, ευελιξία να εφαρμόσουν εξαιρέσεις εκεί που το κόστη είναι δυσανάλογα. Οπότε σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου πραγματικά είναι δυσανάλογο το κόστος υπάρχει δυνατότητα από πλευρά των κρατών μελών να επιλέξουν να δώσουν μια εξαίρεση και άρα να μειώσουν το κόστος χωρίς όμως να μειώσουν το γενικότερο επίπεδο προστασίας. Αυτά ήταν τα τελευταία που είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αρσένης έχει ζητήσει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν είναι νομοθετική πρόταση αυτή για την απαγόρευση των φαρμακευτικών προϊόντων. Έχουμε ήδη υποβάλει τροπολογίες το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιούμε τα φαρμακευτικά προϊόντα που τόσο πολύ χρειαζόμαστε σήμερα, αλλά συγχρόνω να προστατεύουμε και το πόσιμο είδωρ. Πώς δηλαδή θα πετύχουμε το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Αν αυτό επηρεάζει το κόστος, ε, ναι, δεν πρόκειται για ένα φόρο, για ένα τέλος, πρόκειται για μια επένδυση που κάνουμε. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε καλές οικονομικές εξελίξεις ε, στην Ευρώπη γιατί θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης που τόσο πολύ τις χρειαζόμαστε σήμερα. Κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα με τα κράτη-μέλη που είναι αναγκασμένα να τηρήσουν δύσκολες προθεσμίες ή που δεν μπορούν να προετοιμαστούν έγκαιρα. Μα όπως είπε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οδηγία πλαίσιο προβλέπει κάποιες εξαιρέσεις για τις προθεσμίες για οποιοδήποτε χώρα δηλαδή, οποιοδήποτε κράτος μέλος που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προθεσμίες για τις ουσίες αυτές. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιες περιμένουν να είναι οι επιπτώσεις για την απασχόληση με τα επίπεδα αυτά δημοσίων επενδύσεων η οικονομία μας δηλαδή πώς θα αποφεληθεί από την επένδυση αυτή. Και αυτές οι πολύπλευρες επενδύσεις, αν καταφέρουμε δηλαδή να τακτοποιήσουμε το θέμα των τριών αυτών φαρμακευτικών ουσιών ή των παραγόγων τους, θα μπορέσουμε να φιλτράρουμε έτσι και άλλες ουσίες. Είναι δηλαδή μια επένδυση η οποία θα μας βοηθήσει γενικότερα να προστατεύσουμε την υγεία και με πολλούς και άλλους διαφορετικούς τρόπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κρήτον. Ο Ρατάμα τώρα. Ο κύριος Χόλγκερ Κάμερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει και άλλες φορές βλέπουμε ποιες είναι βασικές, τα βασικά στοιχεία της συζήτησης. Ε, μιλάμε για τα, τις τρεις αυτές ε, φαρμακευτικές ουσίες και δεν έχω αμφιβολίες ότι η Επιτροπή έχει δουλέψει με επιστημονικό τρόπο. Αλλά υπάρχουν πολλές νέες πληροφορίες και μελέτες ε, που βάζουν κάποια, θα μπορούσαν τουλάχιστον να θέτουν κάποια ερωτηματικά για το αν αυτές οι τρεις φαρμακευτικές ουσίες πρέπει όντως να είναι στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας. Όταν δεν είναι απολύτως ε, ξεκάθαρα τα πράγματα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε στο πλαίσιο της άσκησης της πολιτικής περιβάλλοντος ε, κατά πόσο ε, θα πρέπει να ε, καταβάλουμε το κόστος και σε τι βαθμό θα πρέπει να καταβάλουμε το κόστος. Και ακούσαμε και αυτά που είπε ο εισηγητής και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις, τα ερωτηματικά τα οποία έχουν τεθεί. Διότι θα πρέπει η κοινωνία, αν αποφασίσει ότι θα πρέπει να βγουν αυτές τις ουσίες από τα ύδατα, θα πρέπει να επιβαρυνθεί και με το κόστος για την αφαίρεση αυτών των ουσιών από τα ύδατα πολύ συχνά είναι και πολύ τοπικού χαρακτήρα ε, αυτές ε, ε, οι επιπτώσεις. Όταν υπάρχει ένα σταθμός βιολογικού καθαρισμού, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι εκεί γύρω ένα προβληματικό σημείο. Θα ήθελα λοιπόν να αποδεχθούμε ότι η συζήτηση είναι ε, τέτοια που μπορούμε να πούμε ότι είναι αμφιλεγόμενο το θέμα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον κίνδυνο, δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε από τον κατάλογο, αλλά νομίζω ότι μπορούν να επιτηρούνται, να είναι αντικείμενο προσεκτικής παρατήρησης και έχουμε και την πολύ απαιτητική οδηγία πλαίσιο για το νερό, Ήδη δηλαδή υπάρχουν προβλήματα για να μπορούν να πληρούνται οι πολύ αυστηρές προϋποθέσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας για να έχουμε μια ισορροπημένη εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Όντως το περιβάλλον κοστίζει, αλλά και ένα κακό περιβάλλον είναι εις βάρος της υγείας. Ο Κάρλος είναι κρίμα που δεν είναι εδώ οι Βρετανοί. Ελπίζω όμως ότι θα το διαβάσουν. Όταν εγώ μελετούσα χημικός μηχανικός, ασχοληθήκαμε και με το θέμα αυτό των υδάτων. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση στη χώρα μου. Αν λοιπόν θέλουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, οι δαπάνες για την Ευρώπη θα είναι τόσο υψηλές που θα ξεπεράσουν κατά πολύ ο οποιοδήποτε όφελος από τα χημικά αυτά. Θα ήταν τρελό δηλαδή οικονομικά να μην σταματήσουμε αυτό που μπορούμε να σταματήσουμε τώρα στην πηγή του. Είναι δηλαδή πολύ πιο οικονομικό, πολύ πιο αποτελεσματικό οικονομικά να το κάνουμε αυτό οι προδιαγραφές ποιότητας που υπάρχουν τώρα είναι βέβαια κάτι καλύτερο από το να περιμένουμε και να δούμε. Γιατί αν περιμένουμε και θα δούμε, περιμένοντας, πολλά, πολλοί θα έχουν κάνει επενδύσεις και μετά θα θέλουν ε, βέβαια κάποια απόδοση. Και αν δεν υπάρχει αυτή η απόδοση, καταλαβαίνετε ότι θα μα έχει κοστίσει πάρα πολύ. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση που οικονομικά το πιο αποτελεσματικό θα ήταν η προστασία του περιβάλλοντο. Αυτό που είναι καλύτερο και για το περιβάλλον δηλαδή συγχρόνω. Τώρα μια πολύ σημαντική πτυχή είναι αυτό που ακούσαμε και πριν για την οδηγία. Ορισμένοι τι κάνουν, υποβάλλουν τροπολογίες και τι λένε. Λένε, μα περιμένετε, υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσεις ανακλάδο. Οι ρυθμίσεις που θα κάνουμε εμείς τώρα δεν θα πρέπει να πειράσουν εκείνες τις ρυθμίσεις. Υπάρχει όμως και το αντίστροφο που λέει ότι αν εντοπίσετε κάτι τώρα μπορεί να μην έχει προβλεφθεί σε άλλε ρυθμίσει, οπότε είναι λογικό να ξεκινήσουμε από εδώ. Αν δηλαδή βρούμε εδώ κάτι και θέλουμε εδώ κάτι να κάνουμε, τότε να αλλάξουμε την όποια ρύθμιση υπάρχει, είτε είναι το ρίτσι, είτε είναι τα βιοκτώνα, είτε οτιδήποτε άλλο. Και αυτό και προσπαθώ και εγώ να κάνω με τις τροπολογίες μου 83 έως 87. Ξέρω ότι ίσως να μην είναι τόσο εύκολο να τις καταλάβει κανείς διαβάζοντάς τις, αλλά Κοιτάξτε, πάρτε δύο λεφτά παραπάνω να τις διαβάσετε και νομίζω ότι θα καταλάβετε. Το νόημα των τροπολογιών αυτών είναι το εξή. Όπου απαιτεί ο κανονισμό αυτό κάποια αλλαγή, θα φροντίσουμε να φτάσουμε και στον αρχικό κανονισμό και να τον αλλάξουμε και αυτόν. Δεν θέλουμε να υπάρχει διαφορά δηλαδή ανάμεσα στου δύο, αλλά θέλουμε να γίνει μια αλλαγή που να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Αυτό που περισσότερο συζητάμε εδώ είναι οι φαρμακευτικές ουσίες βέβαια αλλά και εδώ, τουλάχιστον ε, στις περισσότερες ε, χώρες, πρόκειται για φάρμακα τα οποία δεν συνταγογραφούνται, όπως είναι το τυκλοφενάκ. Στις περισσότερες χώρες που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, δεν χρειάζεται συνταγή. Δίνεται εύκολα και στη Σουηδία, ενώ πριν από μερικά χρόνια δεν ίσχυε αυτό. Τώρα όμως ισχύει. 25 μιλιγκράμμ, ναι. Αν είναι διαφορετικά τα μιλιγράμμα, εντάξει, είναι διαφορετική κατάσταση, γιατί δεν ξέρει κανείς πόσο θα χρησιμοποιήσει ο, κάθε, ο καθένας. Ε, τότε λοιπόν, εφόσον δεν ε, συνταγογραφούνται τέτοια φάρμακα, ε, τα παίρνει εύκολα κανείς και επιτρέπεται και διαφήμιση στην τηλεόραση για τα φάρμακα αυτά. Αν απαιτείται συνταγή, τότε σταματούν οι διαφημίσεις και τότε εξοικονομούμε και χρήματα. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Κράμαρ, πρέπει να μην σπαταλούμε χρήματα για διαφημίσεις ε, τέτοιου είδους. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει νόημα. Σε μερικέ περιπτώσει, εντάξει, μπορεί να μην τα καταφέρουμε να τα απαλείψουμε, αλλά αν μη τι άλλο θα έχουμε εξοικονομήσει τα χρήματα από την διαφήμιση για προϊόντα που θέλουμε να περιορίσουμε. Οπότε και μόνο η απέτηση για συνταγογράφηση βοηθάει το στόχο μας. Προτείνω επίσης την ε, Ιβουπροφένη να τη συμπεριλάβω. υπήρχε πολύ καιρό στον κατάλογο, μετά βγήκε. Νομίζω πάντως ότι υπάρχουν αρκετές ε, μελέτες και αρκετές ανησυχίες για να μπουν σε, στον κατάλογο αυτό που ονομάζουμε κατάλογο επιτήρησης. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να παραμείνουν στα πρότυπα ποιότητα οι ουσίε αυτέ, το γνωρίζετε. Και αν δεν υπάρχει δυνατότητα να το πετύχουμε αυτό, τότε να συζητήσουμε τη συμβαστική πρόταση που προτείνεται. Νομίζω θα ήταν πιο αποτελεσματικό πάντω και οικονομικά και περιβαλλοντικά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή να διατηρηθούν τα πρότυπα ποιότητα περιβάλλοντο. Αυτή είναι η καλύτερη λύση μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Thank you. Um, I take a slightly different view. Um... Σας ευχαριστώ. Έχω μια διαφορετική άποψη κάπως. Εντάξει για τις τροπολογίες που θέλουν να διαγραφούν τα φαρμακευτικά. Και εγώ έχω υποβάλει τέτοιες τροπολογίες. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι απέτυχε να αιτιολογήσει η έκθεση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη συμπερίληψή τους. Και Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν ε, αρκετά στοιχεία γερά, στέρεα, για να συμπεριλαμβάνονται, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Και στηρίζω την άποψη του εισηγητή για να μην ε, βάλουμε μέσα τα πρότυπα ποιότητας, εφόσον δεν υπάρχουν αρκετές επιστημονικές ε, αποδείξεις. Αν δεν υπάρχει αντικειμενική μελέτη, πλήττεται η αξιοπιστία της όλης διαδικασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και άλλη φορά εδώ έχω μιλήσει για το τεράστιο κόστος που έχει η επεξεργασία των υδάτων μετά από τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών. Παρόλα αυτά, ξέρω ότι θα ξανασυζητηθεί τα 27 δις νομίζω ότι είναι δύσκολο να τα δικαιολογήσουμε στον ε, πολίτη. Υπάρχει και ένα επιχείρημα που είναι ενδιαφέρον εδώ που λέει οικονομικά τι είναι το πιο ενδιαφέρον. Ωραία, πολύ λογικό να το σκέφτεται κανείς αυτό και το είπε και ο κύριος Σλέτερ ότι οικονομικά είναι πιο λογικό να περιορίσουμε πράγματα όπως είναι η δικλοφενάκ για να μην ε, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα, να χρειάζεται συνταγογράφηση. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει μελέτη που να έχει γίνει. Δεν υπάρχουν δηλαδή στέρεα στοιχεία επιστημονικά. Μπορεί να έχει ό,τι γνώμη θέλει ο κ. Λίτερ, αλλά να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια άποψη. Γιατί για μένα οικονομικά δεν έχει κανένα νόημα να βάζουμε τον κόσμο να πηγαίνει να παίρνει ραντεβού με τους γιατρούς για να ε, συνταγογραφούν ένα φάρμακο τη στιγμή που ξέρουν εκ των προτέρων ότι αυτό το φάρμακο θα του γράψει ο γιατρός και θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει την επίσκεψη αυτή. Πρέπει σίγουρα να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην ρύθμιση αυτή και άλλες ρυθμίσεις όπως είναι το REACH. Είτε πρόκειται για τα βιοκτώνα, ναι, πρέπει να υπάρχει συνοχή. Αν δεν υπάρχει συνοχή, αυτό πρέπει να διορθωθεί. Έχω υποβάλει διάφορε τροπολογίε όσον αφορά το κατάλογο επιτήρηση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να είναι προσωρινό αυτό ο κατάλογο επιτήρηση, να πρόκειται για επιτήρηση και να πρόκειται για έναν μηχανισμό που θα μπορεί να αφαιρεί ουσίε εφόσον πρέπει από αυτόν. Οι ουσίες που θα υπάρχουν εκεί δεν θα πρέπει να οδηγούν σε προτεραιότητα απαραίτητα. Το είπε και ο εισηγητής Οι ουσίες θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με μια ε, διαφανή διαδικασία, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν μπορεί να βάζεις στον κατάλογο κάτι χωρίς να έχεις διαφανή κριτήρια γιατί το κάνεις. Και αν δεν υπάρξει αυτή η διαφάνεια, δεν χρειάζεται καν να υπάρχει κατάλογος επιτήρησης. Επίσης απογοητεύτηκα που ορισμένοι έχουν υποβάλει τροπολογίες με τις οποίες θέλουν να προσθέσουν και άλλα θέματα πέρα από τον κατάλογο κατά προτεραιότητα ουσιών, επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας. Οι συζητήσεις αυτές δεν βοηθούν πολύ, πιστεύω, παρόλο που τι έχουμε κάνει από την αρχή. Έχουμε καταλήξει σε καθυστερήσει και προβλέπω και άλλε καθυστερήσει με τι τροπολογίε αυτέ, ενώ πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Όπου τώρα σκιώδεις μίλησαν και ο συγητής. Θα δώσω τώρα το λόγο σε άλλους συναδέλφους και να είσαστε παρακαλώ σύντομοι. Δεν θέλω να είμαι αυστηρός, αλλά τουλάχιστον να μην ξοδεύουν πολύ χρόνο. Πίτρε Λίζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σέμπερ για τη δουλειά του, για το σχέδιο που μας παρουσιάζει και το στηρίζω. Ο Κρήτονας έχει δίκιο που λέει ότι η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα από μόνο του και το δίλημα λοιπόν είναι ότι εφόσον βάλουμε ένα τρίτο επίπεδο θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με άλλα ε, άλλες προτάσεις που έχουμε κάνει. Ενώ θα μπορούσαμε από την άλλη να εξοικονομήσουμε και σε κόστος και σε πρώτες ύλες. Αυτό πρέπει να δούμε πώς θα το πετύχουμε. Στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο τελευταία που έχει να κάνει με το PFO. AS και τα PFTs γενικά. Κατά τη γνώμη μου, η νομοθεσία που έχουμε πρέπει να ελεγχθεί γίνονται έλεγχοι στην πηγή, έτσι καλώ απαγορεύονται τα προϊόντα αυτά σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο έρευνας για να προστατεύσουμε το πόσιμο είδωρ, πολύ σημαντικό για την ανθρώπινη υγεία. Οπότε η ερώτησή μου είναι τι γίνεται με τις τιμές 230 φορές περισσότερο είναι ε, οι προδιαγραφέ τη Επιτροπής σε σχέση με το πόσιμο είδωρο. 230 φορές ε, παραπάνω είναι τιμέ. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει ε, το όριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλη η ιδέα για τις ουσίες αυτές σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε τι τιμές βάζουμε και τι νερό θέλουμε να πίνει ο κόσμος. Αυτό πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας όταν καθορίζουμε τις οριακές τιμές. Και για τα φαρμακευτικά φυσικά πρέπει να δούμε τι εναλλακτικέ έχουμε για την για διπλό φενάκι. Όπως λέει και ο Σλέτερ, υπήρξε μια ουσία που βγήκε από την αγορά, κάποια άλλη παραμένει και έχει παρενέργειες όμως. Οπότε τελικά δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο για το πώς θα συμπεριλάβουμε, θα αποκλείσουμε κάποια ουσία. Η υγεία του ανθρώπου βέβαια είναι η προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι βιάστηκε υπερβολικά και θα πρέπει να το ξαναδούμε. Η Κρίστε Κλάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την υποστήριξη που δείχνουν. Ε, εγώ στηρίζω τα όσα είπε ο Ζίμπερ γιατί αυτός ο κατάλογος επιτήρησης είναι καλή ιδέα ο κατάλογος που μας προτείνει η Κομισιόν ε, είναι κάτι το σοβαρό, ωστόσο δεν επηρεάζει σε, το, ποιον κατάλογο υπάρχει κάθε ουσία. Θα πρέπει να υποδεικνύεται πως πρόκειται για μια ουσία που υπάρχει στον τάδε το δίνα κατάλογο. Χρειάζεται ωστόσο επιστημονική βάση. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυθαίρετα, αλλά θα πρέπει να έχουμε επιστημονική βάση. Σίγουρα υπάρχουν ε, ε, κάποιες ουσίες ε, οι οποίες είναι στον κατάλογο, μέταλλα, ορμόνες που βρίσκονται σε μικρή ποσότητα στα ύδατα. Και δεν έχει επιληθεί το θέμα, δηλαδή για μένα δεν πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει επιλύσει το πώς τίθεται τα πρότυπα για τέτοιες ουσίες πολλές φορές ε, ε, επαφείται στα κράτη-μέλη που έχουν ε, τη διακριτική ευχέρεια να ρυθμίσουν ορισμένα θέματα ούτως ώστε να είναι συμβατά με τις οδηγίες και πρέπει να δούμε κατά πόσο τα περιβαλλοντικά πρότυπα καθορίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα να είναι κάτι σαφέστερα προσδιορισμένο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται θα ήθελα να περιγράφουμε και το πώς περιγράφονται οι ουσίες, γιατί ε, το νερό είναι ένα σημαντικό αγαθό και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τα επιστημονικά δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ένα σημείο μόνο είναι αυτό στο οποίο συμφωνούμε, ότι πρέπει το νερό να είναι καθαρό. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο σημείο στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Σε όλα τα άλλα σημεία που άκουσα και από συναδέλφους και από τον Πίτερ Γκάμιλτοφ με κάνουν να σκέφτομαι μα σε ποιο πλανήτη ζούμε. Και φυσικά είναι σωστά αυτά τα οποία ελέγχθησαν ότι θέλουμε καθαρό πόσιμο νερό και ότι πάντοτε χρειάζεται επεξεργασία των υδάτων στο σημείο κατανάλωσης. Βεβαίως, στο τέλος του δικτύου χρειάζεται επεξεργασία. Αλλά η διαχείριση ε, των συνταγογραφούμενων φαρμάκων νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ακούγεται ε, αφελές. Να πούμε σε έναν γυναικολόγο ότι δεν πρέπει να συνταγογραφείτε το α ή το β αντισυλληπτικό. Να πούμε ότι όταν ε, ε, ε, συνταγογραφούνται φάρμακα με δικλοφενάκ είναι κάτι το οποίο αποτελεί, δεν αποτελεί το, το, την λιγότερο κακή λύση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, ε, να υπάρχουν κανόνες και υπάρχουν ε, κανόνες ε, και στο REACH για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πρέπει να είναι αυτά στα οποία υπάρχουν μελέτες και δεν υπάρχει επιβάρυνση από τη συγκέντρωση των ουσιών αυτών των φαρμάκων. νομίζω ότι μπορεί για τη δικλοφενάκ να αγοράσει κανείς τέσσερις ταμπλέτες των 25 μιλιγκράμμ αλλά μπορεί κανείς να πάει σε 10 φαρμακεία και να αγοράσει 10 φορές την ίδια ποσότητα. Επομένως ξέρουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί σε αυτά τα θέματα το μήνυμα που δίνουμε ποιο είναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Ζέμπερ και την Επιτροπή. Θα το πούμε ουσίες προτεραιότητα, θα το πούμε κατάλογος επιτήρηση, δεν με ενδιαφέρει. Θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που επιτηρούμε. Δεν είναι τρόπος αυτός να χειρίσουμε τα πράγματα, έτσι θα κάνουμε πολιτική. Θέλουμε κάποιο αποτέλεσμα τελικά. Όχι να καλυπτόμεθα με φίλο οικεί. Θέλουμε κάτι να ρυθμίσουμε, πώ θα το ρυθμίσουμε. θα μπορούσα να σας απαριθμίσω 100 φάρμακα που μπορεί να θεωρούνται επικίνδυνα. Τα, όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τις χημειοθεραπείες. Όλα αυτά είναι υδροδιαλυτά. Αυτά τα οποία ε, ε, χορηγούνται στον άνθρωπο, είτε ενδοφλεβίως είτε αποστόματος είναι ε, φάρμακα τα οποία έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. το μήνυμα προς τους πολίτες ποιο είναι. Δεν υπάρχει. Από αυτά τα οποία λέτε δεν υπάρχει κανένα μήνυμα προς τους πολίτες. Και δεν υπάρχει και καμία εναλλακτική λύση. Τα ε, ιδιαίτερα επικίνδυνα και τα αεροστατικά φάρμακα της χημειοθεραπείας δεν περιλαμβάνονται εδώ ξέρουμε ότι κάθε φάρμακο είναι δηλητήριο. Όλα τα φάρμακα είναι δηλητήρια. Είναι ένα δηλητήριο που βοηθάει, αλλά σίγουρα έχει και παρενέργειες. Δεν υπάρχουν φάρμακα χωρίς παρενέργειες και έχει παρενέργειες και για το περιβάλλον κάθε φάρμακο. Και εγώ θέλω να απαντήσω στο ερώτημα πώς θα αποφύγουμε αυτές τις παρενέργειες. Και λέει η Επιτροπή ότι θα καταλήξουμε στη λύση που κοστίζει λιγότερο. Τι σημαίνει αυτό? ότι σε κάθε συσκευασία φαρμάκου όταν με πονάει το γόνατο γιατί έπεσα και χτύπησα θα πάρω δικλοφενάκ που όντως παίρνω δικλοφενάκ θα πληρώνω ένα ευρώ παραπάνω στο φάρμακο για να πληρώνω για την καθαρότητα του ύδατος αυτό σημαίνει ε, ε, ε, εξηγήστε μου τι σημαίνει Νομίζω ότι προσπαθούμε να είμαστε ιδιαίτερα κυδαιμονευτικοί, να πούμε «Α, αυτό το φάρμακο δεν μπορείτε να το πάρετε», «Α, αυτά τα αντισυλληπτικά δεν μπορείτε να τα πάρετε», «Όχι, στραδιόλοι, πάρτε κάτι άλλο». Θα κάνουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων, να δούμε ποιο είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Δεν είναι έντιμη αυτή η στάση, αυτό με θυμώνει περισσότερο. Ας πούμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Είναι μια ουσία προτεραιότητα, εμείς όμως δεν κάνουμε τίποτα. Δεν πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε. Απαντήστε μου. Απαντήστε μου σε αυτέ τι Λέει ο Ρίχαρτ Σέβε, θα το αφήσουμε μέχρι το 2026. Γιατί να το αφήσουμε για το 2026. Είναι πολιτική αυτό το να πούμε ότι τα αφήνουμε μέχρι το 2026. Τι να, πούμε ότι δεν θα υπάρχουν αντισυλληπτικά μέσα διόλια, Αποφασίστε τι θα λέμε. Θα τα χρησιμοποιούμε, δεν θα τα χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε καθημερινά ε, κάποια φάρμακα τα οποία εκπέμπουν ε, ουσίες στο περιβάλλον. Και οι αγελάδες ε, επίσης είναι πηγή εκπομπής αερίων που ρηπαίνουν το περιβάλλον και ουσιών που ρηπαίνουν το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Πρέπει να δούμε τι τρόπο ζωής θέλουμε. Θέλουμε ένα τρόπο ζωής που καταστρέφει το περιβάλλον, που επιβαρύνει το περιβάλλον. Μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτόν τον τρόπο ζωής. Όσον αφορά τα φάρμακα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε όχι, δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτόν τον τρόπο ζωής. Εγώ δεν νομίζω ότι μόλις εμείς τα απαγορεύσουμε θα τα πετάξουν στην ε, τουαλέτα ε, ε, οι καταναλωτές και θα σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν αν τα έχουν στην κατοχή τους. νομίζω ότι θα πρέπει να επιλέξουμε μία θέση την οποία να μπορούμε να υπερασπίσουμε χωρίς να ντρεπόμαστε. Και αυτά που άκουσα από τον εισηγητή και αυτά που άκουσα από την Επιτροπή για μένα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βγούμε προς τα έξω και να πούμε ότι αυτό υπερασπιζόμαστε. Μιλάμε για φάρμακα, μιλάμε για καλλιντικά, για αυτά που βάζουμε στο πρόσωπό μας. Είναι προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κόχιν Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυσκολίες για τη φαρμακοβιομηχανία να ακολουθήσει αυτήν την κατεύθυνση και τα πολύ πρακτικά προβλήματα που κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει. Η, κυρία, η συνάδελφος Ροτ Μπέρεντε μας τα επανέλαβε. Ωστόσο, καταρχήν για τις ε, επίμαχες μελέτες. Η πείρα δείχνει πως σπανίως ε, κάνουμε λάθος υπέρ της υγείας ε, και υπέρ του περιβάλλοντος. Όταν κάνουμε λάθος συνήθως ε, γίνεται εις βάρος υγείας και του περιβάλλοντος. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ποιες δυσκολίες έχουμε με διάφορα φαρμακευτικά και φυτογεωνομικά προϊόντα στα λογικού κήπους για να πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Δεύτερον, θα πρέπει στη συνέχεια να συζητήσουμε για προθεσμίες. Βέβαια, 2016 είναι πάρα πολύ μακριά. Οι συνάδελφοι, δεν οι, συνάδελφοι, συμπολίτες, με συγχωρείτε, δεν θα το καταλάβουν αυτό. Ε, είτε είναι ανησυχητικό και πρέπει να δράσουμε μέσα σε μια λογική προθεσμία ή δεν είναι ανησυχητικό. Ε, διαφορετικά ε, υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε μια επικίνδυνη ουσία υποτίθεται ανησυχητική και τις ε, μακρές προθεσμίες. Εντάξει, αν δώσουμε χρόνο να προσαρμοστεί η βιομηχανία, αλλά ένα χρονικό διάστημα το οποίο να είναι λογικό και να είναι και συμβατό με αυτό που περιμένουν οι πολίτες από εμά. Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Ζίμπερ για την, ε, για την ένταξη των τριών φαρμακευτικών ουσιών και κυρίως για τον γλυφοζάτο που σίγουρα έχει γίνει για τα γαλλικά ποτάμια αλλά για μας είναι το πρώτο προϊόν γιατί για την υπόλοιπη ένωση δεν ξέρω είναι το πρώτο ρήπος στα επιφανειακά ύδατα και νομίζω πως είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτού του προϊόντος ε, για να μπορέσουμε να ξέρουμε και να αποφύγουμε τις ε, συνέπειες σε υγειονομικό επίπεδο. Εξάλλου να θυμίσω, όπως έλεγε και ο Κάρλος Λούτερ πριν από λίγο, ότι το ότι λαμβάνεται υπόψη η υγειονομική και περιβαλλοντική επίπτωση έχει οικονομικό αντίκτυπο, αλλά έχει και νόημα από η άποψη οικονομία, εξοικονόμηση για την ανθρωπότητα. Γιατί η αύξηση ορισμένων ασθενειών, των οποίων η υπερβολοντική αιτία έχει πλέον επιστημονικά αποδειχθεί, έχει κόστος για τη δημόσια οικονομία ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε καιρούς ε, τέτοιους δύσκολους είναι ένα στοιχείο διόλου αμεληταίο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλ Χάιντς Φλόρενς. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εγώ θα ήμουν ο τελευταίος που θα μπορούσε να δώσω εδώ μια έξυπνη συμβουλή για το πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε με όλες τις διατάξεις που ήδη έχουμε. Οδηγία για το πόσιμο είδο, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, είδατε και τοπική αυτοδιοίκηση, τι κάνουμε με όλες αυτές τις διατάξεις και τι νοοτροπία έχουμε αναπτύξει, γιατί νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει ε, σε μια νοοτροπία που λέμε ότι κάνουμε, ετοιμάζουμε τις διατάξεις, τις ε, εγκρίνουμε, ε, ακολουθούν οι συζητήσει με το Συμβούλιο και να σας πω και για την οδηγία πλαίσια για το νερό που με είχε απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσπαθήστε, κυρία Λεπάζ, ε, αγαπητοί συνάδελφα, να δείτε τι έχει εφαρμοστεί από όλα αυτά και θα δείτε ε, σε τι άσχημη θέση βρισκόμαστε. Ε, υπάρχει και μια απαγόρευση για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στην Ευρώπη και τα ξέρει η κυρία Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ από τα από τις απαγορευμένες αυτές θέσεις βιολογικών καθαρισμών μπορώ εγώ να σας απαριθμίσω δεκάδες που γνωρίζω ότι υπάρχουν. Και υπάρχουν 50-60 ε, φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία θα βρείτε σε μεγάλη συγκέντρωση και τα χρησιμοποιούν όλοι οι αγρότες και όλες οι μεγάλες εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο και οι αγρότες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα φαρμακευτικά προϊόντα για να παράγουν ασφαλέστερα πατάτες παραδείγματο χάρη. Θα πρέπει να δούμε τι έχουμε αποφασίσει ποια χώρα τα εφαρμόζει, ποια χώρα δεν τα εφαρμόζει. Και στη Γερμανία δεν εφαρμόζονται όλα, μην νομίζετε. Δεν θέλω να κάνω τον κακό και να ψάξω τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι είμαστε αφελείς και ανέντιμοι όσον αφορά την πολιτική των υδάτων. Και η Επιτροπή τα γνωρίζει. Στο ΚΕΛ, στο Ρήνο, οι αρχές δεν είναι σε θέση να ε, πάρουν δείγμα υδάτων από τον Ρήνο. Θα μας πει κανείς ότι ε, σαν κοινοβούλιο είμαστε φεδροί. Καμιά φορά φτάνω στο σημείο να το πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ, Λέω ο Πρόεδρος. Έχουμε κάνει και μια πολύ ε, καλή συζήτηση στο παρελθόν και με τον κύριο Στόιμπερ και μιλήσαμε και για τις προτάσεις της Επιτροπής. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Λίντα Μακάβαν. Yeah, I mean, we have taken long on this. Ναι. Έχουμε όντως καθυστερήσει από τη... σε σχέση με αυτό που είχαμε αρχικά προβλέψει, αλλά νομίζω πως είναι χρήσιμο να ακούμε τα διάφορα επιχειρήματα. Το πρόβλημα μου είναι όμως ότι δεν μπορώ να αποφασίσω και θα ξαναρωτήσω την Κομισιόν, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι πόσο σπουδαίο είναι το πρόβλημα. Γιατί εγώ διαβάζω ξανά και ξανά ότι λείπουν τα στοιχεία. Λείπουν τα στοιχεία και τώρα μιλάω για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι η κλίμακα του μεγέθου του προβλήματο γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Ξέρουμε πω αυτά τα χημικά είναι, ε, δημιουργούν προβλήματα. Δεν ξέρουμε ποιε είναι οι συγκεντρώσει του σε διάφορα κράτη-μέλη. Το ερώτημά μου είναι, αν δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, πώς θα ξέρουμε πώς να χαλάσουμε λύνοντάς το. Ποιο είναι ο αντίκτυπος στην υγεία των ανθρώπων από αυτό το πρόβλημα. Είδαμε κάπως τον αντίκτυπο για τα ψάρια, μα πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν άλλα σοβαρά θέματα στην Επιτροπή Αλληλείας. φαντάζομαι, πιο σημαντικά, φαντάζομαι. Αλλά θα μας πείτε πόσο είναι μεγάλο είναι το πρόβλημα για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Γιατί μας είπατε, το ρωτήσαμε και την περασμένη φορά για να καταλάβουμε ποιο είναι το κόστος. Γιατί είχαμε αυτή την διαφορετικέ εκτιμήσει όσον αφορά τη συμμόρφωση προ αυτέ τι προτάσει, διαφορετικέ εκτιμήσει από εσά, από ε, ε, τι κυβερνήσει κτλ. Όμω είναι πολύ σημαντικό που χαλάμε τα χρήματα, γιατί όπω είπαν και οι συνάδελφοι, τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν σωστά, γιατί είναι δημόσια χρήματα και τη στιγμή που λείπει το δημόσιο χρήμα είναι ακόμη πιο σημαντικό. Δεν έχουμε ακούσει κάτι σχετικό, Εκτό και αν κάτι μα πήρε το Συμβούλιο. Εξακολουθώ λοιπόν να πιστεύω πως δεν έχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες και έπειτα για τη λίστα επιτήρησης βάζονται με κάποια προϊόντα εκεί και θυμηθείτε τι είπε η κυρία Γκέρλινγκ για, τη, για, για τις ουσίες ναι υπάρχει επιστημονική διαδικασία για να μπει κάτι στον κατάλογο αυτό Πώ θα μπουν στον κατάλογο επιτήρηση και τι σημαίνει από τη στιγμή που βρίσκονται στον κατάλογο επιτήρηση, Τι, τι, νόημα έχει για την Κομισιόν αυτό, ο κατάλογο είναι υποχρεωτικό, θα συλλέξουν στοιχεία, θα μείνουν για πέντε χρόνια και πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και έπειτα για το θέμα του ΚΑΛ, για την συνταγογράφηση. Δεν μπορεί νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ποια φάρμακα θα πρέπει να συνταγογραφούνται και ποια όχι. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά που αναφέρατε. Ξέρω όλα και όλα αυτά τα τρία που αναφέρατε. Και γιατί επιλέχθηκαν αυτά και όχι κάποια άλλα και τι σκοπεύει να κάνει στο μέλλον η Κομισιόν για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η κυρία Στρέλα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση ήδη μας δείχνει πως είναι περίπλοκη συζήτηση και αντιφατική, πιο πολύ από ό,τι πιστεύαμε αρχικά και από τη στιγμή που πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, νομίζω πως είναι σημαντικό η συζήτηση να διευρυνθεί όντως και να εμβαθύνουμε στα διάφορα θέματα, γιατί υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και αναπάντητα ερωτήματα όπως υπόθηκε ήδη. Αν λάβουμε υπόψη πως δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία και άρα δεν γνωρίζουμε τη διάσταση του προβλήματος σε καθένα από τα κράτη-μέλη, πράγμα που θα ήταν πολύ σημαντικό για να λάβουμε απόφαση. Και από την άλλη πλευρά, οι τιμές που μας προτείνονται που μας προτείνονται για το στεντιόλ και το δικλοφενάκι είναι ασύμβατες με τις ε, αναλύσεις ε, και τις τεχνολογίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, όπως εξάλλου επιβεβαιώνεται και από μελέτη που μας υπέβαλε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω με τη σειρά μου την Κομισιόν μήπως ε, θεωρεί λογικό σε μια πρώτη φάση οι ουσίες αυτές να συμπεριληφθούν σε ένα κατάλογο επιτήρησης και μόνο μετά, πιο ύστερα, όταν θα έχουμε τα στοιχεία ανάκρατος μέλος και θα γνωρίζουμε, θα έχουμε μάλλον και μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη που θα μας επιτρέπει να περιορίσουμε τις τιμές των ουσιών αυτών, ε, τότε λοιπόν να μπορούμε να τις βάλουμε στο κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας. Γιατί, για παράδειγμα, στη χώρα μου, στην Πορτογαλία, είναι υποχρεωτικό υποχρεωτική επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων φαρμάκων στα φαρμακιά. Αλλά είναι προφανές ότι είναι αδύνατο να ελέγξουμε αν όλοι οι άνθρωποι ε, φροντίζουν το συγκεκριμένο θέμα και ακολουθούν, υπακούν τον κανόνα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ρύθμιση εφόσον πρόκειται για πρακτικές οι οποίες είναι κεκτημένες και περνά πολύς χρόνος για να αλλάξει η συμπεριφορά των πολιτών. Πιστεύω πως πρέπει να ενεργήσουμε, ε, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τη υγεία αλλά να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και ο καλύτερος δρόμος για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθαρό νερό, χρήση, καθαρισμός, όλα αυτά επιβάλλονται για να απαλλάξουμε το νερό από τα δεινά του. Είναι πολύ χρήσιμο για τους ανθρώπους, για τα ζώα. Είναι μια προτεραιότητα που έχουμε και στρατηγική σημασίας προτεραιότητα μάλιστα. Γι' αυτό και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας, τον Σαρζέμπερ, για την ποιότητα ε, του σχεδίου που μας παρουσιάζει έχει καταφέρει να πετύχει δύσκολους συμβιβασμούς, ποιότητας όμως. Οπότε μπράβο του και τον ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που επέδειξε όλο αυτό τον καιρό, που μας άκουσε και έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις μας. Τώρα, ο τρόπος ε, ζωής μας ίσως δεν ευθυγραμμίζεται πάντα με την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να καθίσουμε και να κοιτάξουμε με προσοχή ποια είναι και η οικονομική κατάσταση και η συγκυρία μέσα στην οποία ζούμε σήμερα. Ε, κάποιος το είπε πριν ότι έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς. Εμείς λοιπόν οι ευρωβουλευτές πρέπει να νομοθετήσουμε υπεύθυνα και πρέπει να κοιτάξουμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση των χωρών μας πριν τους επιβάλλουμε νέες υποχρεώσεις για μεγάλα έξοδα. Να μην επαναλάβω όσα έχετε ήδη πει. Δύο σημεία τεχνικά κάπως θέλω να τονίσω. Το πρώτο είναι το εξή. Κάποιες ουσίες, κατά τη γνώμη μου, έχουν θέση όχι τόσο στον κατάλογο ελέγχου χημικών ουσιών, αλλά στον κατάλογο επιτήρησης, γιατί έτσι σε ένα πρώτο στάδιο, αν μη τι άλλο, θα μπορούμε να ελέγχουμε επαρκώς τα προϊόντα αυτά. Το δεύτερο που έχω να προτείνω, και γι' αυτό ο Ρισάρ Ζέμπερ θα λέγω ότι έχει λάβει υπόψη του αυτή την πτυχή, αλλά ίσως όχι ακριβώς έτσι όπως θα το έχω κάνει κι εγώ. Τι εννοώ. Για τον μηχανισμό ε, βάσει του οποίου μπαίνει μια ουσία στον ε, κατάλογο επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας. Υπάρχει μια μεθοδολογία για το πώς μπαίνει σε αυτό τον κατάλογο μια νέα ουσία προτεραιότητας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να προβλέψουμε και μια διαδικασία για να μπορεί μια τέτοια ουσία προτεραιότητας να μπορεί να βγει από τον κατάλογο αυτό, αν αποδειχτεί από κάποια επιστημονική ανεξάρτητη μελέτη ότι δεν έχει λόγο να βρίσκεται σε αυτό το κατάλογο. Ο Ρισάρ ε, Ζέβερ πρότεινε πράγματι να γίνεται μια μελέτη κάθε τέσσερα χρόνια. Μα γιατί να περιμένουμε τέσσερα χρόνια και να μην προβλέψουμε ένα τέτοιο μηχανισμό, ώστε άπαξ και υπάρχει επιστημονική μελέτη ανεξάρτητη που λέει ότι η ουσία ψ δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια βάσει των οποίων βρίσκεται μέσα στο κατάλογο, να μπορεί να βγει από αυτόν. Αυτά είναι λοιπόν τα τεχνικά σημεία που ήθελα να υπογραμμίσω. Είναι πολύ σημαντικό επίσης μαζί να υπολογίσουμε την ισορροπία ε, κόστος-όφελος για το θέμα αυτό πάνω στο οποίο δουλεύουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σλούτα. Σύντομα παρακαλώ. Ε, πολλοί είπαν εδώ ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Ναι, αλλά είναι δυνατόν να τα πουλάμε όλα αυτά τα πράγματα για να μην ξέρουμε τι κάνουμε. Ε, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ανησυχητικό. Και γι' αυτό θελήσαμε να σας ενημερώσουμε και για την σουηδική μελέτη, γιατί προσπάθησαν να φτιάξουν ένα μοντέλο πρόβλεψης, να πούνε δηλαδή ποιες χημικές ουσίες θα έχουν αντίκτυπο και στη συνέχεια ποιες από αυτές τις ουσίες θα έχουν ε, επίπεδα συγκέντρωσης που θα δημιουργούσαν προβλήματα. Οπότε πρώτα είδανε ποια είναι όλα τα χημικά, Πολλά από αυτά τα βγάλανε γιατί είπαν ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουν αντίκτυπο. Κράτησαν 120 υποψήφια από τα οποία ε, βγάλαν 30 που δεν θα είχαν αντίκτυπο και στη συνέχεια το μοντέλο αυτό το σύγκριναν με την πραγματικότητα και ε, σύγκριναν την κατάσταση στην πραγματικότητα και γι' αυτό κατέληξαν σε 15 που είπαν ότι οι συγκεντρώσεις τους είναι αρκετά υψηλέ που άρα είναι ανησυχητικέ, Αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε ποιε είναι ακριβώ οι επιπτώσεις τους ε, πάνω στο νερό, γι' αυτό και φτιάξανε άλλες μελέτες για να δούνε ε, οι συγκεντρώσεις αυτές τι επιπτώσεις θα είχαν στο νερό. Έτσι κι πρέπει κανείς να ακολουθήσει ολόκληρο τον κύκλο ζωής για να μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος. Βρήκανε ένα φαρμακευτικό στοιχείο το οποίο ήταν υψηλότερο στο νερό από ότι στη δόση που ε, καταπίνει με το φάρμακο αυτό ο άνθρωπος. Αυτή η ουσία και στα frog test ε, αποδείχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί διαπιστώθηκε ότι ε, αυτά τα βατράχια, γιατί στα βατράχια έγιναν οι ε, δοκιμές, ε, μπορεί όταν ήταν νεαρά να μην είχαν πρόβλημα, όταν όμως ήταν ενήλικα, τότε φάνηκε ότι υπήρχε το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει κανείς να παρακολουθήσει όλο τον κύκλο ζωής. Λέει και η Ροτ ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Ναι, αυτές οι ουσίες δεν ήταν ουσίες για τις οποίες χρειαζόταν συνταγή ιατρική. Ε, κοιτάξτε, δεν είναι ότι οι Σουηδοί πληρώνονται πέντε φορέ περισσότερο σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν και έχουν λεφτά για να κάνουν τέτοια μελέτη. Πολλέ φορές όταν ε, κάποιος υποφέρει, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα έτσι καλλιώς. Ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη παρέμβαση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κ. Κάτράιτ, εμπειρογνώμων από τον Βρετανικό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Θα ήθελα σύντομα να του δώσω το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας πω ότι εκπροσωπώ την ε, υπηρεσία περιβάλλοντος της Αγγλίας και της Ουαλίας, όχι την Βρετανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά δίνουμε στοιχεία όσον αφορά τα λύματα, έτσι ώστε να φτάσουμε στα ε, προδιαγραφές που ισχύουν και μου ζητήσατε να σας εξηγήσω πώς, στάσαμε, πώς φτάνουμε σε αυτές τις προδιαγραφές. Εκτιμήσαμε λοιπόν 11.000 χιλιόμετρα που έχουμε ποτάμια και ε, Έχουμε τους ε, βιολογικούς καθαρισμούς που λειτουργούν ε, στις όχθες όλων αυτών των ποταμιών. 40% έχουμε ωστόσο επιρροή από τις ηθετικές ορμόνες και 30% έχουμε Ε, το 40% των ποταμιών δεν περνάνε το τεστ των ορμονών και της, ε, της ιστροδιόλης, που είναι η συνθετική ορμόνη. Και φυσικά δεν μπορούμε και να διαχειριστούν τις ε, φυσικές ορμόνες αποτελεσματικά. Το κόστος ε, το οποίο, ε, στο οποίο έχουμε φτάσει είναι 27 με 31 δις λίρες στερλίνες κατά τη μία τριακονταετία. Η χαμηλότερη εκτίμηση σχετιζόταν με την ανάγκη προηγμένης κατεργασίας μέσω της μέσω του ιονισμού. Όμως η... Το μεγαλύτερο κόστος έχει να κάνει με τις βελτιώσεις συμβατικού καθαρισμού των ε, λιμάτων, έτσι ώστε δηλαδή να, καθαρίζεται να ε, καθαρίζονται υπαρκώς τα λίματα. Να σας εξηγήσω επίσης ότι οι πληροφορίες που έχουμε για τις δυνατότητες διαφόρων καταστάσεων καθαρισμού ώστε να φτάσουμε ε, και για να αφαιρέσουμε αυτά τα ιστρογόνα είναι σχετικά μεγάλες. Ανάμεσα στο 2000 και το 2010 ο κλάδος αυτός έκανε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που κόστησε πάνω από 30 εκατομμύρια λίρες και εξέτασε λεπτομεριακά όλους τους συμβατικούς βιολογικούς καθαρισμούς που χρησιμοποιούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και εξετάσαμε πιλωτικά προγράμματα, εξετάσαμε διάφορες προηγμένες τεχνολογίες καθώς και ε, τη, ένα τελευταίας τεχνολογία ε, εργοστάσιο με άνθρακα. Μπορέσαμε να φτάσουμε λοιπόν σε μια καλή κατανόηση του τι μπορούν να επιτύχουν οι διάφορες ε, δυνατότητες κατεργασίες. Αν και η συμβατική κατεργασία μπορεί να φτάσει σε, σε αρκετά καλή αφαίρεση της ιστοδιόλης μέχρι το 72% η εθινολεστραδιόλη που είναι το συνθετικό ε, η συνθετική αντίστοιχη ορμόνη μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μέχρι το 37% ακόμα και με την καλύτερη δυνατή κατεργασία. Μια προηγμένη κατεργασία θα μπορούσε να φτάσει σε αφαίρεση 80 με 90%. Τώρα βέβαια υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο αποτελεσματικό θα ήταν κάτι τέτοιο για να φτάσουμε στις προδιαγραφές για το περιβάλλον. Τώρα, η άλλη, το άλλο σκέλος της προσέγγισης είναι ότι έχουμε εθνικά πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούμε όσον αφορά 3.000 εργοστάσια καθαρισμού, βιολογικού καθαρισμού και εδώ λάβαμε τις εκτιμήσεις για το τι μπορούν να πετύχουν αυτά τα διάφορα εργοστάσια ε, όσον αφορά την ποιότητα της κατεργασίας και το συγκρίναμε με την ροή των ποταμών. Και έτσι έχουμε φτιάξει χάρτες κινδύνου όσον αφορά τις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης αυτών των προδιαγραφών. Κάτι ακόμα που μας επιτρέπει το REACH τώρα είναι να λάβουμε υπόψη την ύπαρξη ουσιών REACH στην ε, αρχή των ποταμών. Πέρα δηλαδή από αυτά τα λίματα τα οποία πέφτουν μέσα στην ε, ροή των ποταμιών. Είδαμε επίση ποιο είναι το ελάχιστο κατεργασία που απαιτείται ώστε να εξασφαλίσουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας που να αντιστοιχεί στι προδιαγραφές. Και έτσι σιγά σιγά φτιάξαμε το κόστος όσον αφορά την προσθήκη περαιτέρω κατεργασία που ήταν απαραίτητη. Για παράδειγμα μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα ύδατα που διατρέχουν κίνδυνο σε 200 περίπου σημεία Ήδη έχουμε την καλύτερη δυνατή κατεργασία ε, ως αποτέλεσμα της οδηγίας περί ε, των ε, ψαριών που ζουν στο γλυκό νερό για να επιτυχθούν δηλαδή τα σωστά επίπεδα περιεκτικότητας σε αμμονία και υπάρχουν κάποιες μικρές βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στα συμβατικά, στους συμβατικούς καθαρισμούς. Ελπίζω πως έτσι θα πήρατε μια ιδέα για το πώς φτάσαμε στο εκτίμηση κόστους κατεργασίας των λιμάτων μας. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που δεν έδωσα το σωστό σας τίτλο στην αρχή. Είσαστε, όπως είπατε, από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος Σουαλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Έγιναν αρκετέ ερωτήσει και προ τον κύριο Κάμελτοφ από την Επιτροπή. Αν θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις μου στις διάφορες ερωτήσεις που μου κάνατε. Πρώτα απ' όλα, υπήρξαν διάφορες ερωτήσεις για το κατά πόσο είναι ένα μέτρο όθησης για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και κατά πόσο είναι μια επένδυση. Για μας είναι και τα δύο. Δηλαδή, αν χειριστούμε το θέμα κατάλληλα, γιατί όπως είπα, είμαστε στην αρχή. Γνωρίζουμε ένα μέρος της τεχνολογίας, δεν γνωρίζουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε εταιρική σχέση για επενδύσεις στον τομέα του ύδατος, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε λύσεις, νέες λύσεις ή λύσεις σε νέους τομείς όπου χρειάζονται τέτοιε λύσει. Αν λοιπόν όλα αυτά τα χειριστούμε κατάλληλα, η ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκός ε, κλάδος επεξεργασίας υδάτων ε, σίγουρα θα γίνει πιο ανταγωνιστικός. Και συγχρόνως θα λυθεί και ένα πρόβλημα που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ενεργεία. Θα δημιουργηθούν δηλαδή θέσεις απασχόλησης και συγχρόνως αν εξάγουμε την τεχνολογία αυτή, επίσης έχουμε να κερδίσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι το φαινόμενο της αστικοποίησης είναι τεράστιο. Όλο και περισσότερο μεγαλώνουν οι πόλεις παντού στην Ευρώπη. Άρα το θέμα αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα πολύ σύντομα τη μια στιγμή την άλλη. Άρα για μας με τον τρόπο αυτό δίνουμε λύσεις και στο περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά και δημιουργούνται νέε θέσει απασχόλησης. Μια άλλη κατηγορία ερωτήσεων είχε να κάνει με τον κατάλογο επιτήρησης. Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στόχος του κατάλογου επιτήρησης δεν είναι να αποφασίσουμε κατά πόσο μείωση είναι επικίνδυνη ή όχι, αλλά να εντοπίσουμε το μέγεθος του προβλήματος, να εκτιμήσουμε το μέγεθο του προβλήματο. Εδώ είναι το θέμα ε, αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα δεν υπάρχει υποχρέωση ελέγχου όσο δεν υπάρχει ουσία στο κατάλογο. Οπότε είναι δύσκολο να έχουμε και στοιχεία δεδομένα από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διανομή προβληματικών, επικίνδυνων ουσιών για το περιβάλλον. Ο κατάλογος επιτήρησης λοιπόν είναι ένας μηχανισμός για να μας βοηθήσει να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Όταν μπει μια ουσία στον κατάλογο επιτήρησης δεν μένει ίσα μένει όσο χρειάζεται μέχρι να εκτιμηθεί δηλαδή κατά πόσο είναι προβληματική αυτή η ουσία ή όχι. Οπότε, κατά τη δικιά μας τη γνώμη, το να μπαίνει μια ουσία στον κατάλογο επιτήρηση σημαίνει ότι μπαίνει ένα, δύο, τρία χρόνια και μετά βγαίνει. Έτσι, σας απαντάω στην ερώτησή σας για το πώς μπορεί να βγει μια ουσία από τον κατάλογο επιτήρησης. Δεν είναι ένα μέρος όπου παρκάρουμε την ουσία και ΜΕΝΙΣΕΙ. Μια άλλη κατηγορία ερωτήσεων ήταν το κατά πόσο καταδικάζουμε κάποιες ουσίε εφόσον ε, τις συμπεριλαμβάνουμε σε επικίνδυνε ουσίε προτεραιότητας. Η απάντησή μου είναι σαφώς όχι. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε δύο ταξινομήσεις ουσιών. Έχουμε τις ουσίες προτεραιότητας και έχουμε και τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας. Οι επικίνδυνες είναι τα T-compounds όπως ξέρουμε και από το REACH και όπου προβλέπεται η εξαφάνισή τους και που προβλέπει 20 χρόνια περίοδο η οδηγία για να αποφασίσουμε πώς θα απαλλαγούμε από την ουσία. Όλες οι άλλες οι ουσίες και οι φαρμακευτικές που αναφέρονται εδώ δεν προτείνονται ως επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητες. Σας το υπενθυμίζω αυτό. Οι ουσίες αυτές Λοιπόν, δεν λέμε ότι πρέπει να καταδικαστούν, αλλά ότι πρέπει η χρήση τους να γίνεται με προσοχή. Τέταρτον. Άλλες ερωτήσεις είχαν να κάνουν με τα αντισυλληπτικά, με τα αντιφλεγμονώδη, με την χημειοθεραπεία, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται δηλαδή στη χημειοθεραπεία. Κοιτάξτε, η Επιτροπή δεν λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις ουσίες. Σαφώς και ο κόσμος τις χρειάζεται και πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στα αντισυλληπτικά, πρέπει να μπορεί να ε, συνεχίζει να παίρνει αντιφλεγμονώδη εφόσον χρειάζονται και βέβαια και πρέπει να έχει πρόσβαση στη χημιοθεραπεία εφόσον η χημιοθεραπεία ενδείκνεται ως κατάλληλη θεραπεία σε έναν ασθενή. Αλλά από την άλλη αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φάρμακο που χρησιμοποιείται είναι το ένα και μοναδικό σωστό. Εμείς λέμε ότι ακριβώς πρέπει να δούμε τι, άλλα, τι άλλες δυνατότητες έχει ένα κράτος να μην στεγογραφεί ένα φάρμακο και ανταυτού να στεγογραφεί ένα άλλο. Αναφέρθηκε και η βουπροφένη. Γιατί δεν είναι στον κατάλογο η βουπροφένη, ενώ είναι η δικλοφενάκη. Είναι γιατί η βουπροφένη ε, αποδομείται πιο εύκολα. Λοιπόν, μήπως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η ουσία αντί για μια άλλη. Δεν θέλουμε βέβαια να μπούμε στα χωράφια των γιατρών, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν αυτή τη δυνατότητα, να αντικαταστήσουν δηλαδή κάποια φάρμακα από κάποια άλλα οι γιατροί κάθε φορά που συνταγογραφούν. Ένα άλλο θέμα ήταν ε, το θέμα των ουσιών που προκύπτουν από τη φυσική διαδικασία στην οδηγία για το είδωρ αναφερόταν η απόσυρση τέτοιων ουσιών που απορρέουν από τόσα καταναλώνουμε, τι τρώμε και τι πούμε και πίνουμε. Το γεγονός ότι είμαστε συγκεντρωμένοι σε μικρές σχετικά επιφάνειες είναι κάτι που δημιουργεί το πρόβλημα. Είναι ο τρόπος ζωής μας. Άρα αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Επίσης υπήρχε το θέμα του αντικτύπου στα λιεύματα. και γενικότερα κατά πόσο γνωρίζουμε την κατανομή των ουσιών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάποιες από τις ουσίες αυτές έχουμε πληροφορίες από λίγες μόνο χώρες μέλη. Έχουμε επιπλέον πληροφορίες από τα όσα γράφονται. Υπάρχουν χώρες μέλη οι οποίες δεν ελέγχουν τις ουσίες αυτές συστηματικά και άλλες που τις ελέγχουν συστηματικά. Όσον αφορά τα λιεύματα, η ανησυχία σας εδώ δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα αποθέματα τα λιευτικά. Ορισμένες από τις ουσίες αυτές επηρεάζουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής των ε, ηχθείων. Δεν είναι γενικά δηλαδή το πρόβλημα των αποθεμάτων, είναι το πρόβλημα το οικολογικό πιο πολύ. Γιατί αν βγάλετε από τον οικολογικό του χώρο το ψάρι, τότε κάτι λείπει στο οικοσύστημα και τότε μπορεί να δημιουργηθούν ε, άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ρωτήσατε και για την εφαρμογή. Υπήρξε πρόσφατα μια έκθεση για την ε, εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά τα αστικά λίματα. Τις επόμενες εβδομάδες θα δημοσιευθεί μια μεγάλη έκθεση για την εφαρμογή της ε, οδηγίας πλαίσιο για το είδωρ. Οπότε κύριε Φλόρενς, κοιτάξτε την. Σίγουρα θα υπάρξει και ευκαιρία να τη συζητήσουμε. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη εφαρμογή των όσων έχουμε ήδη. Φυσικά και πρέπει να εφαρμόζονται και φυσικά και πρέπει να ενσωματώνονται καλύτερα στη γενικότερη και να εντάσσονται καλύτερα στη γενική πολιτική. Αλλά έχει να κάνει όντω με την εφαρμογή και συγχρόνω αξιολογούμε ποιε άλλε ουσίε δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον. Τέλος, κάποιες παρατηρήσεις για το κόστος. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά όλα όσα είπατε. Και εκπρόσωπος της Αγγλίας και της Ουαλίας, ε, της υπηρεσίας περιβάλλοντος δηλαδή. Το κόστος προϋποθέτει ότι όλα ο στόχος μας είναι η τελική λύση και γι' αυτό μιλάμε για το ανώτατο κόστος πάντα. Εμείς στη δικιά μας έκθεση αντικτύπου μεταξύ άλλων έχουμε πει 11 με 18 ε, το χρόνο κατά κεφαλή ως κόστος. Άκουσα τι είπατε για το επιπλέον κόστος στην Αγγλία για τα 20 χρόνια, για το πακέτο ολόκληρο. Για μένα είμαστε στα 25 με 30 κατά κεφαλή το χρόνο. Έτσι. Αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς τι μέτρα πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα έχουμε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, κάτι που πρέπει να αποφασιστεί από τα κράτη-μέλη. Οπότε τελικά καταλήγουμε σε αντίστοιχα στοιχεία πρέπει να σας πω με αυτά που έχει ανακοινώσει και η Γερμανία. 10 με 30 ευρώ δηλαδή τελικά είναι το εύρος για την ε, επεξεργασία που θέλουμε. Και τέλος, αν υπάρχουν επιπλέον ωφέλη, ναι, αν εφαρμόσετε τέτοιου είδους επεξεργασία, τότε απαλλάσσεστε και από ένα σωρό άλλα χημικά, άλλες χημικές ουσίες που βρίσκονται και ανοιχνεύονται στο είδωρ. Άρα γλιτώνεται και από άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα και λυπάμαι αν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ και δίνουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ζέβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Ευχαριστώ και την Επιτροπή και τον εμπειρογνώμονα από την Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πόσο σημαντικό ήταν το να ασχοληθούμε και άλλη μια φορά σήμερα με αυτό το θέμα, γιατί και η Επιτροπή χρειάστηκε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις και ακόμη παραμένουν πολλές ερωτήσεις που δεν έχουν επιληθεί και στις διαπραγματεύσεις μας εξάλλου. Θέλουμε να έχουμε όσο δυνατόν καθαρότερα ύδατα και για τις μελλοντικέ γενιές στο μέλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας κοινό μας στόχος και ήδη έχουμε επιτύχει πολλά και θέλουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω λεπτομερώς για όλα όσα αναφέρθηκαν. Το προτινόμενο πλαίσιο από την Επιτροπή και αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα κινούνται προς την κατεύθυνση που και εμείς όλοι θα θέλαμε και νομίζω ότι όλοι μας ε, αυτό θα θέλαμε, να επιτύχουμε δηλαδή ε, την καλή χημική κατάσταση του ύδατος. Όσον αφορά τώρα τα νομικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε και τις λεπτομέρειες επ' αυτού, νομίζω ότι μπορούμε στις διαπραγματεύσεις να τα διευκρινίσουμε. Βλέποντας τις τροπολογίες, πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο κοντά από ό,τι θα πίστευε κανείς. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε και τι θα κάνουμε με τις φαρμακευτικές ουσίες. Με την οδηγία για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα έχουμε ένα καλό εργαλείο για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να προσθέτουμε περαιτέρω διατάξεις και νομίζω με βάση τα κριτήρια τα οποία θα καταρτίζει η Επιτροπή αυτό μπορούμε να το κάνουμε και η Επιτροπή έχει συνεργαστεί πολύ καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Ε, παρόλα όσα έχουμε ακούσει και σήμερα και σε προηγούμενες συζητήσεις με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο φαίνεται ότι δεν έχει φτάσει ακόμη η στιγμή ε, η κατάλληλη για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε ε, αυτά τα πρότυπα και ίσως γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε για να θεσπιστούν αργότερα. Όλα αυτά τα μέτρα σχετίζονται με απαιτήσει ελέγχου σε επίπεδο περιφερειών και σε τοπικό επίπεδο στα κράτη-μέλη και αυτό είναι ιδιαίτερα ε, δαπανηρό. Ε, πιστεύω ότι και τα άμεσα και τα έμεσα αποτελέσματα και επιπτώσεις αυτών των διατάξεων που έχουμε σήμερα σε αυτή την έκθεση θα είναι συνολικά ε, θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει παράλληλα με αυτά τα οποία συζητήθηκαν για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν ότι εδώ έχουμε μια πολιτική για τη διαχείριση των πόρων. Η διαχείριση των υδάτων είναι ένας στόχος και για την Ευρώπη του 2020 και μιλάμε για ε, ένα πολύ σημαντικό πόρο ε, που θα πρέπει να διαχειριστούμε καταλήλως θα συνεννοηθούμε με τους σκιώδεις συζητητές και νομίζω ότι θα μπορέσουν οι πολιτικές ομάδες να καταλήξουν σε μια κοινή θέση. Δεν είναι τόσο διαφορετικές οι θέσεις μας για να μπορέσουμε να πιέσουμε και το Συμβούλιο να κάνει κάποια ε, κίνηση προς τη δική μας κατεύθυνση ούτε ώστε να καταλήξουμε σε αυτό που όπως σας είπα είναι η σωστή χημική ποιότητα του ύδατος για τώρα και για τις μελλοντικέ γενιές. Νομίζω αυτά θα είναι τα αντικείμενα των μελλοντικών μας συζητήσεων και με χαρά θα περιμένω τις συζητήσεις με τους σκιώδεις συζητητές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν με την έκθεση αυτή κυρία Ζέντα. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 17 Νοεμβρίου είναι 7 ε, Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου στις 12 ε, και προβλέπεται η ψηφοφορία της ε, έκθεσης στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Περνάμε στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης τώρα. Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη, την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου και από πλευρά μου να συγχαρώ τη συνάδελφο Κρίστα Κλάς για τη θέση την οποία ανέλαβε από σήμερα. Συγχαρητήρια. Και Περνάω στην ε, ενωσιακή πολιτική προστασία. Είδαμε ότι στην αρχή της συνεδρίασής μας μια συνάδελφος μίλησε για πλημμύρες, ε, για καταιγίδε, μεγάλες βροχοπτώσεις που έγιναν στη χώρα της. Αν σας θυμίσω εγώ ως Ιταλία, μάλιστα ως Ιταλίδα, χτες μόλις ε, είχαμε την επέτειο 46 ετών από την τρομερή καταστροφή και τις πλημμύρες που έγιναν το 1936 ή ε, στη Φλωρεντία. Ε, τεράστιες ζημιές υπέστη η καλλιτεχνική κληρονομιά μας που είναι και κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ε, ε, θυμήσαμε για τους άγγελους της Λάσπης. χιλιάδες κόσμος που ήρθε από όχι μόνο από την Ιταλία τότε αλλά από ολόκληρο τον κόσμο για να σώσουν αυτή την εξαιρετική και πολιτιστική κληρονομιά που είναι όπως επαναλαμβάνω κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας και για να βοηθήσουν τον πληθυσμό που πραγματικά είχε ισοπεδωθεί τότε. Πιστεύω πως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε αυτά τα γεγονότα γιατί από την μνήμη των όσων έχουν συμβεί στο παρελθόν και που δυστυχώς συνεχίζει να συμβαίνει και με τις κλιματικές αλλαγές βλέπουμε πως έχουμε να αντιμετωπίσουμε δραματικές ε, φυσικές καταστροφές όλο και πιο συχνά Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη βούληση και την πεποίθηση ότι πρέπει και να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα, γνωρίζοντας πως ήδη έχουμε μεγάλη εμπειρία, τεράστια εμπειρία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και από την οποία να, να, να, να πάρουμε το κουράγιο και την βούληση να κάνουμε καλύτερα και περισσότερα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, διότι συμμετείχαν με πολλές τροπολογίες 226 για την ακρίβεια. Τροπολογίες οι οποίες ε, πιστεύω θα μας επιτρέψουν να δουλέψουμε εξαιρετικά και να δώσουμε μια περαιτέρω όθηση, να ορίσουμε καλύτερα την πρόταση ψηφίσματος και να έχουμε ένα πραγματικά αποτελεσματικό μέσο. Για να απολοποιήσουμε την ανάλυση και να είμαι σύντομη, γιατί πιστεύω ότι το σημαντικότερο στοιχείο σήμερα είναι ε, να ακούσω, να είμαι ανοιχτή στους συναδέλφους από τις διάφορες χώρες και από τις διάφορες πολιτικές οικογένειες. Πιστεύω λοιπόν πως οι τροπολογίες θα μπορούσαν να μοιραστούν σε τρεις μεγάλες ομάδες, τρεις βασικές ομάδες. Στην πρώτη θα τοποθετούσα τις τροπολογίες που στόχο έχουν να αποσαφηνίσουν την σύνταξη της ε, νομοθετικής πρότασης. Τροπολογίες δηλαδή που θέλουν να αποφύγουν ε, την σύγχυση και τις παρεξηγήσεις. Για να συνεννοούμαστε, εδώ βάζω όλες τις τροπολογίες όπου δίνεται προσοχή σε έννοιες όπως η εθνική κυριαρχία, η τοπική η περιφερειακή διάσταση, οι κλιματικές αλλαγές κτλ. κτλ. Αυτές οι τροπολογίες δεν αλλάζουν ε, την φύση της νομοθεσίας, ούτε το νόημά της. Όμως πιστεύω πως βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η κατεύθυνση των προθέσεών μας και ποιες είναι οι ανησυχίες μας. Στη δεύτερη ομάδα ε, έχω τοποθετήσει τις τροπολογίες που στόχο έχουν να αποδυναμώσουν κάπως την πρόταση να αποδυναμώσουν λοιπόν την πρόταση και είναι εκείνες οι τροπολογίες που κατά βάση εγώ θέλω να τις λάβω υπόψη γιατί είναι τροπολογίες που κρύβουν ανησυχίες οι οποίες είναι απόλυτα θεμητές και ελπίζω πως θα καταφέρουμε στη συνέχιση των εργασιών μας ε, όταν θα προχωρήσουμε εις βάθος και στις πρακτικές πτυχές θα καταφέρουμε να τις ξεπεράσουμε. Ξεπερνώντα δε αυτέ τι ανησυχίε, είμαι πεπισμένη ότι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την πρόταση. Εν γέννη, αυτές οι τροπολογίες φαίνεται να προτείνω ότι το σημερινό status quo αρκεί και ότι δεν χρειάζεται αυτό το ποιοτικό άλμα που τελικά όμως όλοι μας επιθυμούμε. Επίσης υπάρχει αυτή η έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, πρέπει να παρεμβαίνει σε κάτι που είναι ευθύνη των κρατών μελών. Τέλος έχουμε μια τρίτη ομάδα ε, τροπολογιών που στόχο έχουν το αντίθετο, που θέλουν να ενισχύσουν την πρόταση της Κομισιόν, να την σπρώξουν λίγο περισσότερο δηλαδή. Μεταξύ αυτών τοποθετώ εκείνους που θέλουν να πούμε περισσότερη χρηματοδότηση για τις μεταφορές και μεγαλύτερη προσοχή στην προετοιμασία. Επιπλέον, ωστόσο, αναλύοντας όλες τις τροπολογίες, ήθελα να πω ότι αν γέννη ε, η συμφωνία είναι εφικτή, γιατί υπάρχει σύγκληση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την πρόταση αυτή. Δεν θέλουμε να μεταφέρουμε εξουσίε περαιτέρω στην Επιτροπή, ούτε θέλουμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να εκμεταλλευτούν την καλή βούληση άλλων. Π.χ. Μιλώντας για τα εθελοντικά, την εθελοντική συγκέντρωση μέσων, ε, να ανταποκριθούμε στις φυσικές καταστροφές πιο αποτελεσματικά, να σώσουμε περισσότερες ζωές και να αλληλοβοηθηθούμε. Στόχος είναι δηλαδή εμείς ως Κοινοβούλιο να συμφωνήσουμε σε μια υπεύθυνη θέση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις διάφορες ευαισθησίες και τις ανησυχίες όλων. Γνωρίζουμε αλλά θέλω να το επαναλάβω, πως οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν περισσότερη Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Είναι ένα από τα λίγα θέματα που οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν περισσότερη Ευρώπη. Όταν λοιπόν γίνεται ένα αίτημα περισσότερε Ευρώπη από πλευρά των συμπολιτών μα, δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να του κάνουμε να αισθανθούν πω ε, η Ευρώπη είναι το κοινό μα σπίτι και ότι έχει ένα φιλικό πρόσωπο και αλληλέγγυο πρόσωπο. Και κατά την άποψή μου αυτό ο μηχανισμό αντιπροσωπεύει και μια μεγάλη ευκαιρία για να εξοικονομήσουμε χρήματα αντιμετωπίζοντα τι ε, καταστροφέ που είναι όλο και πιο ε, επαναλαμβανόμενε, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε εκείνο το είδος καταστροφών που δεν είναι πολύ πιθανό να συμβούν αλλά έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο για τις οποίες ένα μόνο κράτος μέλος από μόνο του είναι πιο δύσκολο να είναι προετοιμασμένο ε, να είναι προετοιμασμένο δεν έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα αίτημα αλληλεγγύης, ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και εγώ ειλικρινά ελπίζω πως το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορέσει να βρει μια συμφωνία για αυτή την μικρό, το μικρό αλλά ταυτόχρονα και μεγάλο βήμα μπροστά ώστε οι ζωές των συμπολιτών μας να είναι πιο ασφαλείς. Τούτο λεχθέντος. Να πω ότι άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, να πω ότι είμαι εδώ για να ακούσω περαιτέρω προτάσεις και ενδεχομένως να απαντήσω και σε ερωτήσεις τους. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Γκαρντίνη. Η ε, κυρία Τέλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Καρντίνη για την έκθεσή της, που πιστεύω ότι έχει μια ρεαλιστική αντιμετώπιση για να βελτιωθούν οι στόχοι του μηχανισμού. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες, δεν θα τις σχολιάσω βέβαια όλες, Θέλω όμως να πω δύο λόγια για ορισμένες από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και που νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντες. Οι τροπολογία του κύριο Σουβένς όσον αφορά το διεθνές σύστημα. Κατά τη γνώμη μου αξίζει τον κόπο να διατηρηθεί. Βλέπω ότι οι προτάσεις αυτές μπορεί να πρέπει να περάσουν από έλεγχο στο Συμβούλιο, αλλά είναι ενδιαφέρουσες πάντως όσον αφορά την ανθρωπιστική πτυχή. Η κυρία Στρέλα επίσης έχει υποβάλει κάποιες ενδιαφέρουσες τροπολογίες, ιδιαίτερα για τον τρόπο που θα λειτουργεί το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Όποιος δεν έχει έρθει σε επαφή με κέντρα που κάνουν αυτή τη δουλειά, του συστήνω να πάνε γιατί αξίζει τον κόπο. Οι τροπολογίε τη κυρία Χάση επίση είναι ενδιαφέρουσε και του κυρίου Ρώση είναι επικοδομητικέ, παρόλο που υπάρχει και ένα θέμα που ελπίζω ότι τελικά δεν θα περάσει. Και αυτό είναι το να γίνονται όλα σε θελοντική βάση. Ορισμένα στοιχεία της πρότασης μπορούν να μείνουν προαιρετικά, όπως η συλλογή πόρων, για παράδειγμα, αλλά πιστεύω ότι η συμμετοχή στον μηχανισμό γενικά αν ναι, είναι σε θελοντική βάση θα ήταν σφάλμα. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος ε, στέλνει πληροφορίες, ενημερώνει, οργανώνει, οπότε δεν πρέπει να αφήνεται σε οποιονδήποτε μπορεί να θέλει να βοηθήσει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είναι σε θελοντική βάση συμμετοχή στο μηχανισμό, γιατί τότε αποσταθεροποιείται ο μηχανισμός. Ως σκιώδη εισηγητές θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Κάποια πράγματα θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο. Σίγουρα η θέση μας πρέπει να παραμείνει ισχυρή, κυρίως για το υποχρεωτικό των σχεδίων και της μη θελοντικής βάσης για τη συμμετοχή στον μηχανισμό. Η κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ. Ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Στρέλα, αλλά ήθελα να δω και τα έγγραφά μου πρώτα. Δίνω όμως το λόγο στην κυρία Στρέλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι φυσικές καταστροφές αυξάνουν σε συχνότητα. αλλά και σε ένταση. Όπως πολύ πρόσφατα απέδειξε ο κυκλώνας Σάντι που έδωσε ένα χτύπημα καταστροφικό στις Ηνωμένε Πολιτείες, στην Αιτή και άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό έχει να κάνει με τις ε, κλιματικές αλλαγές, με την ε, αστικοποίηση, αλλά και με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στις πολιτικές πρόληψεις αλλά και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διαχείρισης των καταστροφών και ε, να δοθεί μια ολοκληρωμένη απάντηση. Και αυτό ακριβώς στοχεύει να κάνει αυτού τη η πρόταση. Εμείς ε, ως ε, ομάδα των σοσιαλιστών υποβάλαμε διάφορες προτάσεις τροπολογίας με στόχο να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ανταποκριθούμε φυσικά στις προσδοκίες των πολιτών που κατά βάση είναι υπέρ της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πολιτικής, πολιτικής προστασίας που θα οδηγεί στη χαρτογράφηση των περιοχών κινδύνου αλλά και στη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε απάντηση στις καταστροφές. Και γι' αυτό και υποστηρίζουμε ότι οι δράσεις πρόληψης πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο μια απογραφή αλλά και μια χαρτογράφηση των κινδύνων ε, καθώς και μια έγκριση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων που θα πρέπει να λάβει υπόψη τις αξιολογήσεις ανάλυσης κινδύνου περιφερειακού και τοπικού επίπεδου. Και μάλιστα αυτά τα σχέδια να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2014. Όσον αφορά την ε, ανάπτυξη ικανοτήτων ανταπόκρισης σε επίπεδο ένωσης, ε, έχουμε την εντύπωση ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται εκεί οι ικανότητες της οριζόντιας ώστε να μπορούν να ανταποντήσουν ε, σε επίπεδο ε, πρόληψης, ε, υλικοτεχνικής υποστήριξης, ε, ακόμα και όταν πρόκειται για τις καταστροφές μικρής πιθανότητας αλλά υψηλού αντικτύπου έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα αποθεματικό αεροπορικών μέσων για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, πράγμα το οποίο αιτιολογείται Θεωρούμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να προβλέψουμε κίνητρα για τα κρατημέλη που θελοντικά διαθέτουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας στεναρής ευρωπαϊκής δυνατότητας απάντησης. Προτείνουμε λοιπόν την, α, την αύξηση διατήρησης των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής της Ένωσης για ανταπόκριση στα στις φυσικές καταστροφές και αύξηση 90% για το σύνολο των διαθέσιμων ποσών ώστε να εξαλειφθούν οι ελλείψεις, να καλυφθούν οι ελλείψεις. Θεωρούμε επίσης πως η αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο τα κράτη, αλλά και ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να μειώσουν ε, τις επενδύσεις τους σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό δηλαδή τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης και το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας. Επίση, θεωρούμε πως είναι σημαντικό να εγγυηθούμε την ενίσχυση της διαφάνειας της εθνικής στρατηγικής προετοιμασίας και γι' αυτό ε, προτείνουμε ε, Κομισιόν να στηρίξει την δημιουργία ε, εθελοντικών προαιρετικών εκτιμήσεων κινδύνου που γίνονται από τα κράτη-μέλη, την ανταλλαγή των πρακτικών, αλλά με βάση κριτήρια προκαθορισμένα, ώστε να μπορούν να γίνουν και συστάσεις για να ενισχυθεί το επίπεδο προετοιμασίας της Ένωσης. Όπως ε, παρουσιάστηκαν 263 τροπολογίες, θεωρούμε πως θα ήταν σκόπιμο η συγκήτρια να υποβάλει κάποιες προτάσεις συμβιβαστικές και φυσικά είμαστε στη διάθεσή της ώστε να αναλύσουμε και να συμβάλλουμε ε, έτσι ώστε τελική εργασία και τελική πρόταση να είναι μια πρόταση ε, συνεκτική ε, και να αντιστοιχεί στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να, καταρχήν να συγχαρώ τη συνάδελφο Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη για την έκθεσή της, αλλά και επειδή συστηματικοποίησε τα θέματα τα οποία διακυβεύονται όταν μιλάμε για αυτό τον ε, μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Ήδη υπόθηκε ότι οι κλιματικές αλλαγές βρίσκονται στη, ε, στην ρίζα και στην προέλευση της νομοθετικής αυτής πρότασης γιατί, ε, και, γιατί ο αριθμός των φυσικών καταστροφών έχει αυξηθεί καθώς και η ένταση αυτών. Οι φυσικές καταστροφές λέγονται φυσικές καταστροφές, ωστόσο πολλές από αυτές έχουν να κάνουν με τις ε, κλιματικές αλλαγές ε, με ανθρωπογενείς ε, παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον και επηρεάζεται όχι μόνο ο κόσμος αλλά και η κληρονομιά, η ηλικία αλλά και η πολιτιστική. Θα έχουμε χρόνο για να το συζητήσουμε να συζητήσουμε και συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ θα ήθελα μόνο να αναφέρω τρεις ιδέες κλειδιά σε σχέση με τη θέση της ομάδας μου και που βρίσκονται στην ε, βάση των τροπολογιών που υπέβαλα. Ε, πρώτο θέμα είναι ότι προφανώς πέρα από τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και τις εσωτερικές τους υποχρεώσεις γιατί έχει να κάνει αυτό με τη δική τους επικράτεια, τους πολίτες τους κτλ. Είναι, υπάρχουν και αμοιβέ υποχρεώσεις σε σχέση με άλλες ε, χώρες. Πέρα λοιπόν από αυτές τις υποχρεώσεις που ήδη υπάρχουν για κάθε κράτος μέλος, πιστεύουμε πως ο συντονισμός σε περίπτωση καταστροφών δεν μπορεί να γίνεται ad hoc βιαστικά και μετά από τα συμβάντα. Γι' αυτό και θεωρούμε πως είναι απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα συντονισμός μέσων και μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ανταπόκριση και απάντηση. Είναι προφανές πως πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αλληλοβοήθειας αλλά και συμβατότητα και ολοκλήρωση των σχεδίων ε, κινδύνου και η αξιολόγηση αυτών των κινδύνων. Η ε, πρόληψη φυσικά είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για ένα θέμα ε, τόσο βευρύ και αν θέλουμε να μιλήσουμε για το ποια μπορεί να είναι η πρόληψη για κάθε ένα από αυτά τα θέματα, αυτές τις περιπτώσεις μάλλον ε, φυσικής καταστροφής, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Αλλά είναι προφανές πως η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά το ίδιο σημαντική είναι και η ολοκλήρωση, η ολοκληρωμένη απάντηση. Από αυτή την άποψη, όπως είπα, χωρίς να επηρεάζεται η κυριαρχία των κρατών μελών, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να τα συντονίσει αυτά, ώστε να μπορέσουν και τα κράτη-μέλη πιο αποτελεσματικά να δράσουν, τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Ένας αλληλέγγυος μηχανισμός, λοιπόν, για αυτόν συζητάμε και με αυτό συμφωνούμε, θα πρέπει να είναι ένας μηχανισμός ε, κατεξοχήν πολιτικού χαρακτήρα και ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, σε περίπτωση που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν πολιτικά μέσα αλλά και στρατιωτικά θα πρέπει αυτό να γίνει αλλά θα πρέπει να, να είναι σίγουρο πως αυτό θα γίνει πάντοτε ε, σύμφωνα με τις αρχές ανθρωπικής βοήθειας και ότι οποιαδήποτε κλίση, επίκληση μάλλον με στρατιωτικών δυνάμεων για να βοηθήσουν σε πολιτικού χαρακτήρα ε, ε αποστολές πρέπει να γίνεται μετά από αίτημα των κρατικών αρχών και όχι με αυτόνομη ενέργεια, αυτενέργεια των στρατιωτικών αρχών. Γι' αυτό και έχουμε υποβάλει την τροπολογία 211 που στηρίζει αυτή την έννοια. Δηλαδή πάντοτε να υπήρχε πολιτικός έλεγχος όσον αφορά την συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων. Σας ευχαριστώ. Eu <laughs> Ναι, δεν μίλησα και 10 λεπτά. 10 λεπτά δείχνει το χρονόμετρο, αλλά δεν μίλησα 10 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα πάντα. Φυσικά και πρέπει να μιλήσουμε για την πρόληψη, για το συντονισμό και για την ανταλλαγή των πρακτικών. Όμως θέλω να σας πω ότι η ομάδα μας, CCR, στηρίζει τη γενική ιδέα της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ε, τέτοιων κινδύνων. Οι ανησυχίες μας ε, πάντως και οι τροπολογίες μας έχουν να κάνουν με την επικουρικότητα τουλάχιστον όταν πρόκειται για προσπάθειες οι οποίες πάνε πέρα από τις αρμοδιότητες του άρθρου 196 της συνθήκης. Για παράδειγμα, η απέτηση, ε, τα σχέδια ε, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να πρέπει να τα μοιραζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θέλουμε να αποφασίσουμε κάτι το οποίο να συμμορφώνεται πλήρως με τις συνθήκες. Και δεν θέλουμε 100% ε, να είναι κοινέ οι δράσει αυτέ, γιατί στο μέλλον κάποιε χώρε μπορεί να θέλουν να κάνουν τι δικέ του επενδύσει στον τομέα αυτό τη πολιτική ε, προστασία. Είναι πολύ ανησυχητικό, κατά τη γνώμη μας, να υπάρχει τέτοια αύξηση στον προπολογισμό για τον τομέα αυτόν έτσι όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, ε, χαιρόμαστε για την πρόταση όσο αυτή παραμένει αναλογική, λογική και στα πλαίσια της συνθήκης και εφόσον προσφέρει κάποια προστιθέμενη αξία, κάτι παραπάνω. Να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικαταστήσει τις υποχρώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη. Βεβαίως θα είμαστε παρόντες για συμβαστικές τροπολογίες και ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον συνάδελφο Πέταλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η εισηγήτρια γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση και γνωρίζει τι απαιτείται να γίνει, όπως επίσης γνωρίζει και τι είναι εφικτό να γίνει. Και γι' αυτό τη συγχαίρω για την έκθεσή της που είναι πολύ καλή. Η κλιματική αλλαγή δείχνει ότι ε, οι διατάξεις που αφορούν την πολιτική προστασία γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικές και οι ανάγκε μας είναι όλο και μεγαλύτερες. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προπολογισμού και δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε συνεχώς αυξήσεις των διαθέσιμων πόρων. Θα πρέπει λοιπόν με ορθολογικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση χωρίς ε, να δημιουργήσουμε γραφειοκρατικά προγράμματα για τα οποία θα χρειαζόταν ακόμη πιο ακριβή χρηματοδότηση σε μια εποχή περιορισμένων πόρων. Θα ήθελα να σχολιάσω την πρόταση που αφορά το 46. Θα σας πω για ποια τροπολογία μιλάω. Για την τροπολογία 259 οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα και γι' αυτό θα πρέπει σύμφωνα με τις αρχές μας και σύμφωνα με τις αξίες μας να δίνουμε βοήθεια και στις χώρες που είναι υποψήφιες χώρες ή ε, χώρες που δεν βρίσκονται τώρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε και το μέσο προενταξιακής βοήθειας, όπως επίσης και το μέτρο για την πολιτική γειτονίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζέμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη για την έκθεσή της, γιατί αυτός ο τομέας της καταπολέμησης των ε, φυσικών καταστροφών ε, είναι ένας τομέας όπου για την Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό να εργαζόμαστε από κοινού. Και αν δούμε τις δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκό πρόσωπο σε αυτό τον τομέα. Δεν υπάρχουν σύνορα στις φυσικές καταστροφές και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ευρωπαϊκή συνεργασία. Βεβαίως την ε, αρμοδιότητα έχουν τα κράτη-μέλη και η δική μας ε, πολιτική ομάδα επιμένει ότι χρειάζεται ευρωπαϊκός συντονισμός και καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η πολιτική πίεση είναι μεγάλη σε τέτοια θέματα και μπορούμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένα σημεία. Νομίζω ότι πολύ σωστά συμπληρώνει η συγγήτρια την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή ήθελε μόνο ε, πράξεις ε, εφαρμοστικές, ενώ η Ελιζαβέτα Γκαρντίνη μιλά και για πράξεις κατεξουσιοδότηση πιστεύω ότι χρειαζόμαστε σαφώς καθορισμένα κριτήρια και δεν θα πρέπει να περιμένουμε να υποβάλει την πρόταση η Επιτροπή για να μπορέσουμε μετά να ζητήσουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω. Καλό θα ήταν από τώρα να καθορίσουμε το τι είναι για μας σημαντικό και από την αρχή να ακολουθήσουμε την πορεία την οποία θέλουμε και όχι να επιρρύψουμε την ευθύνη στην Επιτροπή αν κάτι δεν έχει γίνει αργότερα. Πάντω είναι πολύ καλή η πρόταση γενικά και ελπίζω ότι θα μπορέσει να τύχει υψηλή πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Ρίχαρντ Ζέμπα και δίνουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ο κύριο Ντά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας και την εισηγητριά σας, αλλά και τους άλλους ευρωβουλευτές που στηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εμείς πιστεύουμε ότι οι περισσότερες από τις προτινόμενες τροπολογίες είναι θετικές και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την πρότασή μας. Η στήριξη αυτή για μας είναι πάρα πολύ σημαντική για μας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει για ένα τέτοιο θέμα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι συμφωνείτε με τις απόψεις μας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί ε, ευθυγραμμίζεται απόλυτα και με τις απόψεις των ε, πολιτών. Από τα πρόσφατα ευρωβαρόμετρα φαίνεται ότι οι πολίτες μας στηρίζουν αυτές τις προτάσεις. Είναι επίσης σημαντικό για μας γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να μας βοηθήσετε να αντιμετωπίσουμε τις τάσεις που υπάρχουν στο Συμβούλιο για να περιορίσουν την πρόταση αυτή. Συνεπώς προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σας και στην ενεργό στήριξή σας στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Έρχομαι τώρα σε μερικά συγκεκριμένα θέματα που θίξατε. Πρώτα απ' όλα, ε, συμφωνώ και εγώ με αυτό που λέει η κυρία Γαρδίνη, ότι το status quo σίγουρα δεν φτάνει. Αυτή είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεν φτάνει γιατί οι κίνδυνοι αυξάνονται χάρη και στις κλιματικές αλλαγές σε ένα μεγάλο βαθμό. Έπειτα υπάρχουν και νέοι κίνδυνοι που αναδύονται και που μέχρι τώρα δεν έχουμε αναλύσει αρκετά. Πρέπει να προετοιμαστούμε και για αυτούς. Για παράδειγμα, ε, ηλιακές καταγίδες. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο και να προετοιμαστούμε. Και είναι κάτι που βέβαια δεν μπορεί να γίνει από κάθε χώρα χωριστά από μόνη της. Πρέπει μαζί να βάλουμε τις δυνάμεις μας. Όπως επίσης και οι κρίσεις που έχουμε μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει με τρόπο εντελώς απρόβλεπτο πολλές χώρες στον, στον πλανήτη μας. Το τελευταίο παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών ε, δείχνει κατάφορα, πιστεύω, ότι χρειάζεται δράση και ότι χρειάζεται δράση τώρα. Μάλιστα, ε, συχνά ε, το πρόβλημα προκύπτει όταν έχουμε οικονομικές δυσκολίες. Και αυτό είναι ένας παραπάνω λόγος για τον οποίο χρειάζεται συνεργασία και να βρεθούν τρόποι ώστε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και τις καταστροφές με όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό τρόπο που να μην κοστίζει πολλά. Πολλοί επικεντρώθηκαν στην πρόληψη, ότι χρειάζεται περισσότερη πρόληψη, περισσότερη οργάνωση και σχεδιασμός έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να καλύπτουμε ημέν τα κενά των άλλων. Τώρα εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος για το εξή. Τίποτα από τόσα προτείνει η Επιτροπή δεν θέλει να αντικαταστήσει τα κράτη-μέλη. Αντίθετα, η νομοθεσία αυτή υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη ποιε είναι οι δικέ του βασικέ ευθύνε στον τομέα τη πολιτική προστασία. Δεν θέλουμε να του αφαιρέσουμε καμία από αυτέ τι αρμοδιότητε και ευθύνε. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει η επικουρικότητα και ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν όσο γίνεται περισσότερε ευθύνε και αρμοδιότητε σε αυτά <clears throat> τα θέματα και τα συστήματά τους αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα. Εχειρόμαστε επίσης που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να εμείνει στην θέση του. Όπως και η κυρία Τέιλορ, θέλω και εγώ να υπογραμμίσω το θέμα της εθελοντικής συμμετοχής ε, στις ικανότητες των κρατών μελών και γενικότερα στο μηχανισμό. Αυτό που θέλουμε είναι να πετύχουμε μια καλή ισορροπία, δηλαδή να ενισχύσουμε την προβλεψιμότητα της συνεργασίας από τη μια και από την άλλη να παραμείνουν οι ευθύνε και αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εθελοντική δράση. Άρα ισορροπία ψάχνουμε, μια ισορροπία που να μας επιτρέψει να ε, ανεβάσουμε τον πύχη στον τομέα της συνεργασίας στην πολιτική προστασία. Είναι πολύ σημαντικό για μας να περάσουμε σε μία προσέγγιση που να βασίζεται περισσότερο στην πρόληψη των κινδύνων παρά στη διαχείρισή τους. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι ελαστική για την διάρθρωση και για το πώς στην πράξη τίθεται σε εφαρμογή κάτι τέτοιο. Πάντως, η ανταλλαγή πληροφοριών είναι σίγουρα ένα πολύ βασικό σημείο κίνησης. Πρέπει να ξέρουμε πόσες χώρες ε, μέλη αξιολογούν ε, προβλέπουν τους κινδύνους και σε τι βαθμό. Έτσι θα καταλάβουμε καλύτερα τι κινδύνους έχουμε μπροστά μας. Τώρα για το θέμα της εθελοντικής συμμετοχής. Το οικονομικό σκέλος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ιδέα αυτής της εθελοντικής ε, συμμετοχής είναι κάτι που θέλουν όλες οι χώρες. Είναι κεκτημένο πια στο Συμβούλιο. Και αυτό που εδώ μπορούμε να υπογραμμίσουμε είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Χρειάζονται κίνητρα προκειμένου τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια, στην κοινή ικανότητα. Και τα οικονομικά φυσικά είναι στρατηγική σημασίας. Και αυτό γιατί είναι κάτι που σίγουρα κοστίζει και είναι ένα κόστος το οποίο κανονικά δεν συμπεριλαμβάνεται στον ε, προπολογισμό πολιτικής προστασίας των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη δηλαδή από το δικό τους ε, τον προπολογισμό, έχουν χρήματα για να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές και τα λοιπά στο δικιά τους την επικράτεια, αλλά δεν λαμβάνουν ποτέ υπόψη το κόστος στην περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσουν άλλες χώρες μέλη με τις δικές τους καταστροφές. Αν λοιπόν θέλετε ένα αποτελεσματικό σύστημα συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών, ο μόνος τρόπος για να το πετύχετε είναι το κόστος μεταφοράς να το συμπεριλάβετε στο ευρωπαϊκό κόστος τέλος, ο κίνδυνος ε, ηθικής ζημίας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά. Φυσικά δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, συστήματα τα οποία να πηγαίνουν πέρα από την ε, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Χρειάζεται όμως και πάλι μια ισορροπία. Έχουμε συμπεριλάβει εδώ προβλέψεις για περισσότερη διαφάνεια από πλευρά των κρατών μελών όσον αφορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και το πώς ε, προβλέπουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους αυτούς. Έπειτα υπήρξε και το θέμα του peer review που τον έφεραν κάποιοι από εσά. Πολύ καλός τρόπος για να υπάρχει διαφάνεια μεταξύ των χωρών μελών. Τέλος, για την ευρωπαϊκή χρηματοδοτούμενη ικανότητα έχουμε το low probability high impact risks. Είναι κίνδυνοι δηλαδή μεγάλη αλλά μικρής πιθανότητας που σήμερα δεν ε, μελετώνται τόσο πολύ. Για 27 χώρες δύσκολο η καθεμία να επενδύσει από μόνη της σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό και θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία, να γίνει δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε πώς θα μοιραστεί το κόστος μεταξύ μας. Αυτά είναι τα κύρια θέματα που είχα να σας αναφέρω. Και κάτι ακόμα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Είναι το ένα. Και το δεύτερο, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Τέιλορ. Δηλαδή, το κέντρο ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικό και όσοι από εσά θέλετε να το επισκεφτείτε μπορείτε να το κάνετε. Θα ήταν πράγματι χρήσιμο να υπάρξει μια σύντομη συνάντηση εκεί, γιατί μια τέτοια εμπειρία βοηθάει τον κόσμο να καταλάβει περισσότερο στην πράξη τι δουλειά γίνεται και ποιε είναι στην πράξη οι ανάγκε που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο κέντρο. Η συγκίτρια τώρα, τελευταία μιλήτρια, η κυρία Καρδίνη. Σα ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. σα ευχαριστώ για τη συζήτηση που ήταν πολύ θετική. Νομίζω πω ε, όλε οι παρεμβάσει ήταν σημαντικές και συμφωνώ με όλες. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που είπε η Κομισιόν, ισορροπία. Νομίζω πως πρέπει να βρούμε αυτή την, ε, ε, ε, αυτό το σημείο ισορροπίας όπου όλοι να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι πέρα από κάποιες ευαισθησίες και κάποιες ανησυχίες είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Δουλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Είμαι πολύ αισιόδοξη λοιπόν και ελπίζω πως σύντομα θα μπορέσουμε να βρούμε σύγκληση. Δέχομαι την πρόσκληση της ε, κυρίας Εστρέλα και των υπολείπων συναδέλφων για να μπορέσουμε να ε, φτιάξουμε συμβιβαστικές και πιστεύω πως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με κάποιες διμερείς ε, συναντήσεις για να εμβαθύνουμε σε κάποια θέματα και να βρούμε και τρόπο να προχωρήσουμε. Όπως ε, με τη συνάδελφα Ναρόσμπαχ, ας πούμε, παρά τις ε, ανησυχίες της, ε, συμφωνούμε, νομίζω, επί της βάσης για το ποιος είναι ο τελικός στόχος που θέλουμε να πετύχουμε. Άρα θα μπορέσουμε και αυτή τη φορά, νομίζω, να τα βρούμε να θυμηθούμε ότι με βάση αυτά που είδαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγο ένα χρόνο στην Ιαπωνία, τις εικόνες ε, του τυφώνα Σάντι ε, και, και ακόμα και μεγάλες χώρες υπερδυνάμεις κατάλαβαν πως πολλές φορές δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους ε, να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές και κυρίως διαπίστωσαν και συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν και αυτοί φτάσανε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να σκεφτούμε το απίστευτο πια. Και άρα πρέπει να έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Είναι προφανέ πω το status quo δεν μπορεί να είναι το σημείο άφηξη, αλλά το σημείο αφετηρία από το οποίο θα πρέπει να κινηθούμε πια. Και από το Συμβούλιο έφτασαν και έγιναν μεγάλα βήματα μπροστά, ακόμα και αν η Κομισιόν εξακολουθεί να πιστεύει πως το κοινοβούλιο είναι το, ο οίκος όλων των πολιτών και άρα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τις προσδοκίες και τις απαιτήσει των συμπολιτών μας πέρα από τις θεσμικές ανάγκες με τις οποίες ασχολούνται συνήθως οι κυβερνήσεις και βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Σας ευχαριστώ λοιπόν ακόμα μια φορά. Θα προχωρήσουμε με τη συνεργάτη μα στην δουλειά για να φτάσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην ε, έκθεση. Είδαμε μάλιστα φέτος το καλοκαίρι κάποια παραδείγματα που λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά, κάποια πιλωτικά προγράμματα όπου υπήρξε δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις καλοκαιρινές πυρκαγιές. Ξέρουμε ότι ορισμένα από αυτά τα πιλωτικά προγράμματα τελειώνουν φέτος και δεν θα μπορούμε να, δηλαδή να αφήσουμε ακάλυπτες τις ε, περιοχές μας. Σίγουρα σχεδόν του χρόνου θα έχουμε ένα κενό σε αυτή την ε, δυνατότητα ανταπόκρισης. Γι' αυτό και πρέπει να δουλέψουμε σωστά αλλά και γρήγορα. Αυτό θα ήθελα και πιστεύω αυτό θέλουν και οι συμπολίτε μας στην ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκαρντίνη στην Επιτροπή θα γίνει η ψηφοφορία 28-29 Νοεμβρίου και είναι μια έκθεση στην οποία θα συνεργαστείτε με την Επιτροπή ΔΕΔΕ. Το επόμενο σημείο είναι η τροποποίηση της Οδηγίας 2536 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Μη σας φαίνεται απίθανο, είναι κάτι το οποίο επιδιώκουμε και θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Άνια Βάισκερμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την καλή συνεργασία που είχαμε σε πολλά σημεία. 83 κοινέ τροπολογίες ε, έχουμε μαζί προσπαθώντας να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής. Σε πολλά σημεία υπήρχε συμφωνία. Υπάρχουν δέκα τροπολογίες στις οποίες μπορούμε να συντομεύσουμε την ψηφοφορία γιατί συγκεντρώσαμε πολλές ε, τροπολογίες ε, σε συμβιβαστικές ε, συγκεντρωτικές τροπολογίες. Και η Γκουε, παρότι είχε ψηφίσει μια τροπολογία, την απέσυρε και τελικά συμπεριλήφθηκε στην συμβαστική τροπολογία. Θα προσπαθήσω εν συντομία να σας παρουσιάσω αυτές τις εργασίες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την γραμματεία. Η συνάδελφος Ρωμάνο, ε, ε, καθώς και τους συνεργάτες μου, θέλω όλους να τους ευχαριστήσω γιατί πιστεύω ότι με τη βοήθειά τους καταφέραμε πολλά ε, δύσκολα σημεία. Υπάρχει ένα σημείο που αφορά τις γλωσσικές απαιτήσει εδώ έχουμε τις τροπολογίες 1, 9 και 10, όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροπολογίες που αφορούσαν αυτά τα θέματα. θέλαμε η Επιτροπή Υγείας να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς όσον αφορά τις γλωσσικές απαιτήσει στον τομέα της υγείας. Μερικές φορές είναι πραγματικά απαραίτητο να υπάρχουν τέτοιες ε, γλωσσικές γνώσεις γιατί είναι ε, επαγγέλματα τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με τους ασθενείς και γι' αυτό ε, χρειάζονται γλωσσικές απαιτήσει και μιλάμε για το επίπεδο C1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου γνώσεων. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι απαιτούνται γλωσσικές εξετάσεις που θα ε, διασφαλίζουν το επίπεδο γνώσεων της γλώσσας στο C1. Βελτιώσαμε τις προτάσεις της Επιτροπής, πιστεύω, και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να βρούμε μια λύση και για τις χώρες όπως το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, όπου υπάρχουν ε, πολλές επίσημες γλώσσες. Και στη συμβαστική μας τροπολογία έχουμε πει ότι θα πρέπει να ε, εξετάζεται η γλώσσα της περιοχής στην οποία πρόκειται να εργαστεί ε, ο εν λόγω πολίτης. Ε, βαλονικά στην Βαλονία, γαλλικά στη Βαλονία, φλαμανδικά στην, ε, στη Φλάνδρα. Και νομίζω ότι αυτές οι τροπολογίες 1, 9 και 10 μπορούν να υποστηριχθούν από όλες τις ομάδες. Στην 9 και 10 νομίζω ότι οι φιλελεύθεροι και ε, οι οι κομμουνιστές, οι Λίνκε δεν συμφωνούν για την 9 και 10. Υπάρχουν ε, κάποια θέματα που αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ε, του ετούντος. Ε, θα πρέπει να δίδεται επαγγελματικό διαβατήριο ή επαγγελματική ταυτότητα κατόπιν αιτήσεως του συγκεκριμένου πολίτη ή ε, κατόπιν αιτήσεως ε, του ε, επαγγελματικού συλλόγου. Αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν να ελέγχονται και μετά από ένα χρόνο για να ελέγχεται το αν συνεχίζουν να ισχύουν αυτές οι πληροφορίες. Όλα αυτά τα κάνουμε γιατί έχουμε κατά νου την ασφάλεια των ασθενών. Η Επιτροπή είχε προτείνει δύο χρόνια, νομίζω το status quo ήταν ένα χρόνος και αυτό προτιμούσαν οι σοσιαλδημοκράτες και το ECR να παραμείνει δηλαδή το ένα έτος. Όσον αφορά την ε, έκδοση άδεια, εδώ έχουμε τις συμβαστικές τροπολογίες 5 και 6. Νομίζω ότι είναι τροπολογίες ε, που μπορούν να γίνουν αποδεκτές από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, θα ήταν, κίνδυνος, θα ήταν επικίνδυνο το να μην υπάρχουν αυτές οι εγκρίσεις, να μην δίδονται εγκρίσεις και να θεωρείται ότι δίδεται η έγκριση μετά από κάποια προθεσμία πραξίας. Έχει μπει και κάποια προθεσμία εδώ, δηλαδή τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν επαρκές χρονικό διάστημα για να εξετάσουν τα επαγγελματικά προσόντα και να ζητήσουν ε, και νέες πληροφορίες από το κράτος μέλος προέλευσης αν το θεωρούν απαραίτητο. Και δεν θέλουμε στη συνέχεια το κράτος μέλος υποδοχής να απορρίψει μία αίτηση για να αποφύγει την σιωπηρή έγκρισή της. Θα πρέπει να δούμε αν θα δίδεται μία προσωρινή έγκριση σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την κινητικότητα. Όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών, εδώ συμφωνήσαμε ότι τα κράτη-μέλη για το προσωπικό υγείας μπορούν να επιτρέπουν αυτά τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών. Η δική μου τροπολογία μάλλον ε, προχωρούσε περισσότερο από όσο ήθελαν οι άλλες πολιτικές ομάδες και υπάρχουν οι τροπολογίες των συναδέλφων Περίλιο Φερέρα που μάλλον ε, κινούνται προς την κατεύθυνση του να ε, απορρίπτεται η αίτηση χωρίς να αποκλείεται όμως κάποια αίτηση της. Πιστεύω ότι είναι καλή η συμβαστική τροπολογία στην οποία έχουμε καταλήξει με αμοιβαίες παραχωρήσεις. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα στο οποίο νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Το θέμα των ε, νοσηλευτών ε, και νοσοκόμων είναι η συγκεντρωτική τροπολογία 8 που επίσης ε, έχει υποστήριξη από πολλές πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Από όλες τις πολιτικές ομάδες υπευλήθησαν τροπολογίες για το σημείο αυτό. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτό δεν είναι καθαρά γερμανικό θέμα, δεν είναι κάτι που συζητείται μόνο στη Γερμανία. Η πρόταση να γίνουν από 10-12 τα έτη για την πρόσβαση στο επάγγελμα προτάθηκε και από άλλα από τις κάτω χώρες, παραδείγματος χάρη στις στις κάτω χώρες Υπάρχει ένα ε, πολύ ποιοτικό σύστημα κατάρτισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των ε, νοσηλευτών και δεν απαιτούνται 12 έτη. Και για τη Μάλτα υπάρχει κάτι αντίστοιχο και για την Ουγγαρία και για την Σλοβακία. Και στην Αυστρία και στο Λουξεμβούργο υπάρχει ε, διτή εκπαίδευση. Στην Ευρώπη Υπάρχουν δύο οδοί που οδηγούν στο πτυχίο νοσηλευτού. Ε, η μία οδός μιλά για δωδεκαετή εκπαίδευση και η άλλη οδός μιλά για δεκαετή εκπαίδευση και επαγγελματική εξειδικευμένη σχολή Και σε αυτό το διτό σύστημα που αναφέρθηκε ότι έχουν και κάποιες ε, άλλες χώρες, ε, είναι, έχουμε σύστημα ε, με θεωρία και πρακτική άσκηση παράλληλα στο πλαίσιο των σπουδών. Στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση που είναι διαφορετική, δεν λέω ότι δεν είναι εξίσου καλή, λέω ότι είναι απλώς διαφορετική. Εκεί είναι χωριστή η θεωρία από την πρακτική και η πρακτική άσκηση ακολουθεί τη θεωρητική εκπαίδευση. Στα περισσότερα κράτη-μέλη τουλάχιστον. Πάντως και οι δύο οδοί μας οδηγούν στο στόχο μας και αυτή η διτή εκπαίδευση, δηλαδή θεωρία και πράξη παράλληλα, είναι πολύ επιτυχημένη εκπαίδευση στην ε, Αυστρία και στο Λουξεμβούργο και η ανεργία των νέων είναι χαμηλή και πιστεύω ότι είναι θετική αυτή η δυτή εκπαίδευση που ακολουθείτε και είναι ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσαν να δεχθούν και άλλες χώρες. Κατά τη γνώμη μου η Επιτροπή κάνει ένα λάθος θέλει να βελτιώσει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και επικεντρώνει την προσοχή της αποκλειστικά στη σχολική εκπαίδευση. Θα έπρεπε να ασχοληθεί με την κατάρτιση γενικότερα, πράγμα το οποίο δεν κάνει. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η Επιτροπή ασχολείται μόνο με τη σχολική εκπαίδευση. Και νομίζω ότι και στο παράρτημα ε, που υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις φαίνεται ότι η Επιτροπή ασχολείται μόνο με τη σχολική εκπαίδευση. Δεν θέλησαν ούτε η Επιτροπή ούτε οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι να το βάλουμε μέσα στην έκθεσή μας. Πάντως υπάρχουν χώρες ε, που εμπίπτουν σε αυτή την ε, περίπτωση ε, και θεωρώ ότι περιορίζεται η κινητικότητα. Εμείς ε, αναζητήσαμε ένα συμβιβασμό στις ε, συγκεντρωτικές μας τροπολογίες. Ναι κύριε Πρόεδρε δεν θα μακρηγορήσω, τελειώνω. Στη συμβιβαστική μας τροπολογία λέμε τουλάχιστον 10 χρόνια, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υποβαθμίζουμε το σύστημα που έχουν κάποια κράτη-μέλη, λέμε τουλάχιστον 10 χρόνια και σε μία πρόταση το λέμε ξεκάθαρα ότι σε ορισμένε χώρες ε, ε, το σύστημα είναι διαφορετικό και έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι επιπλέον. Και είδα και τις τροπολογίες της κυρίας Ροτ Μπέρεντ για ελάχιστη ηλικία 16 ετών κατά την ε, έναρξη της ε, πρακτικής άσκησης, ώστε να μην έχουμε ε, πολύ νεαρά παιδιά σε αυτή την κατάρτιση. Και υπάρχει και η παράγραφος 3, στην οποία παραπέμπουμε, για να προβλέπουμε πόσες ώρες πρακτικής άσκησης και θεωρίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά τμήματα. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν μια έκκληση προς όλους τους συναδέλφους να υποστηρίξουν αυτή τη συγκεντρωτική τροπολογία υπαριθμών 8 γιατί δεν υποβαθμίζουμε την εκπαίδευση που ήδη υπάρχει παγιωμένη και επιτυχή σε πολλά κράτη-μέλη και επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν αυτό το οποίο ε, ε, επιθυμούν. Ανέφερε τα κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικά συστήματα και θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή ΙΜΚΟ και στην, επόμενη συζήτησή μας ε, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία για άλλη μια φορά δεν συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία με τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά συμφωνήσαμε στα βασικά σημεία και νομίζω ότι στην ψηφοφορία αύριο θα μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ροτ Μπέρεντιν, Μάριο Πιρέλο, Παρανόβα, Γιανακουδάκης. Φερέιρα, Αναρόσπαχ και Έντιτ Εστρέλα. Ο Ρίχαρτ Ζέμπερ, Καρλ Χάιντς Φλόρενς, Πέτερ Λίζε και Ντάγμαρ Ροτ Μπέρεντ. Και Κοθίν Λεπάς και κλείνει ο κατάλογος των αγοριτών. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να είναι σύντομοι. Γιατί έχουμε και άλλη μια έκθεση της κυρίας Βέστλουντ. Μάριο Περίλιο έχει το λόγο ο σκιώδης συζητητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την ε, τόσο καλή δουλειά που έχει κάνει και που έχει καταφέρει να βρει κάποιες συμβαστικές ε, λύσεις συμβαστικές λύσεις με τις οποίες οι πολιτικές ομάδες γενικά συμφωνούν. Παραμένει βέβαια το θέμα που έχει να κάνει με την γενική εκπαίδευση των ε, νοσηλευτών. Πολλές τροπολογίες θέλουν να παραμείνει 10 χρόνια. Να πρέπει κανείς δηλαδή να έχει πάει σχολείο 10 χρόνια πριν να μπορέσει να σπουδάσει νοσηλευτής. Η γενική εκπαίδευση να αυξηθεί στα 12 χρόνια, αυτό αιτιολογείται, λένε, εξαιτία των ε, εξελίξεων που έχουμε στον ε, νοσηλευτικό τομέα γενικά και τον ιατρικό τομέα. Διότι πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνολογίες κάποιος, κάπως πιο περίπλοκες από ό,τι κατά το παρελθόν. Οι προϋποθέσεις καθορίστηκαν το 1977, πριν από 30 χρόνια δηλαδή. Σε αυτά τα 30 χρόνια οι περισσότερες χώρες, 24 στις 27 τουλάχιστον, είπαν ότι πρέπει οι ελάχιστες απαιτήσει να προσαρμοστούν για να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στις σπουδές νοσηλευτή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι μετά από 12 χρόνια γενική εκπαίδευση μπορούν να σπουδάσουν οι νοσηλευτές και ότι αυτό ευθυγραμμίζεται με την ε, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για παράδειγμα που προτείνει ως ελάχιστη ηλικία τα 18 χρόνια για να μπορεί κανείς να σπουδάσει νοσηλευτής νοσοκόμος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι πολύ βασικά και έχουν τεράστιες ευθύνες οι νοσηλευτές, συνεπώς χρειάζεται η αναγκαία οριμότητα και ικανότητες για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ασθενών. Καλό λοιπόν τους συναδέρφους να σκεφτούν, να σκεφτούν πολύ και καλά για να αποφύγουμε να καταλήξουμε σε μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων. Οι χώρες που έχουν μειώσει την ηλικία έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες Πρέπει όμως να έχουμε μία Ευρώπη όπου να μπορούν όλοι να συνεπάρχουν. Η ε, κύριε, Γερκοδάκη, ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βάσπεργκερ για τη δουλειά της που προσπάθησε να πετύχει συμβιβασμούς για τα πιο βασικά ζητήματα όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. Το μήνυμα πρέπει να παραμείνει το ίδιο ότι πρώτα απ' όλα προέχει η ασφάλεια των ασθενών. Ιδίω όταν μιλάμε για τα επαγγέλματα υγεία. Τώρα, εκ μέρου τη ε, Άλντε, θέλω να σα πω ότι συμφωνώ με τι βασικέ τροπολογίε 7 και 9 που αναφέρονται στα γλωσσικά προσόντα, τι επαγγελματικέ ταυτότητε και τον αποκλεισμό από την μερική πρόσβαση των επαγγελμάτων ε, που έχουν να κάνουν ε, με επαφή με τους ασθενείς. Θέλουμε να διευκρινίσουμε επίσης τις θέσει μας όσον αφορά στους τροπολογίες 8 με 10 ή 10 τροποποιεί ε, τον γλωσσικό έλεγχο που καταρχήν είχε να κάνει με όλα τα επαγγέλματα και είχε να κάνει με την αμοιβαία αναγνώριση και όχι ειδικά με ε, τα ιατρικά επαγγέλματα. Η Επιτροπή λέει ότι πρέπει να είναι αναλογικές ε, οι εξετάσεις για τα γλωσσικά προσόντα, κάτι το οποίο μας φαίνεται λογικό. Η διατύπωση Επίσης για Consolidated είναι αντιφατική πιστεύουμε, διότι μιλάει για την αναλογικότητα, συγχρόνως όμως βάζει πολύ υψηλά επίπεδα γλωσσικών γνώσεων, το C1 ε, επίπεδο, που είναι πολύ ψηλό. Δεν έχει νόημα λοιπόν να έχουμε αυτές τις δύο αρχές στην ίδια διάταξη, γιατί έτσι τελικά επιβαρύνονται υπερβολικά με εξετάσεις άτομα τα οποία μάλιστα δεν έρχονται σε επαφή με ασθενείς. Πρέπει να ζητάμε επίπεδο C1 για έναν ο οποίος ασχολείται με τη συντήρηση γεωργικών μηχανμάτων. Έχει νόημα αυτό. Για την τροπολογία 8 συζητήσαμε ήδη εκτενώς. Και εδώ επαναλαμβάνω τη στήριξή μου στην απέτηση για 12 χρόνια γενική εκπαίδευση όταν πρόκειται για νοσοκόμους πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ε, ίδιο επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα αρχής, ισοτιμίας, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας των ασθενών. Δεν παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας εδώ, εφόσον χώρες όπως η Γερμανία που έχει δύο εκπαιδευτικά συστήματα μπορεί να τα διατηρήσει σε εθνικό επίπεδο. Αλλά όταν πρόκειται για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να χρειάζεται ε, μια ελάχιστη προδιαγραφή γενικής ε, σχολικής εκπαίδευσης που να απαιτεί και οριμότητα για αυτούς που θα γίνουν νοσοκόμοι και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο τελικά των ιατρικών υπηρεσιών. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες οργανώσεις νοσοκόμων θέλουν να διατηρήσουμε την απέτηση των 12 ετών και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσοκόμων κλπ. όπως και οι οργανώσεις ε, φοιτητών νοσοκόμων. Θέλω να σας πω ότι στην αρχή προσπαθούσα να καταλάβω όχι μόνο τι συμβαίνει στη Γερμανία, αλλά και αλλού. Γιατί υπάρχουν ε, αυτές, ε, αυτοί δύο δρόμοι σπουδών. Τελικά κατάλαβα ότι κάποιες από, κάποιοι από τους νοσοκόμους δεν έχουν καν απολυτήριο λυκείου δεν έχουν ολοκληρώσει την μέση εκπαίδευση και δεν θα μπορούν να αναβαθμιστούν με bachelor και master με κάνει να σκέφτομαι το ότι δεν είμαστε σε μια κατάσταση που χρειαζόμαστε πηγόντως νοσοκόμους αν κάποιες χώρες θέλουν τόσο γρήγορα να φτιάχνουν νοσοκόμους, υπονομεύουν τις ε, σπουδές που κάνουν σε άλλες χώρες οι αντίστοιχοι επαγγελματίες. Διαφωνούμε λοιπόν με την μείωση στα 10 χρόνια και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα στραβό μήνυμα που θα στείλει η Επιτροπή μας στην ΙΜΚΟ και θα υπονομεύσει επίσης και την ασφάλεια των ασθενών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τον κύκλο των σκιωδών εισηγητών. Εσείς είστε ε, αντικαταστάτης, δεν είστε σκιώδης εισηγήτρια. Σας είπα ότι έχουμε και τη την συζήτηση για την έκθεση Westlund και γι' αυτό δεν θα ήθελα να σας δώσω τόσο πολύ χρόνο. Παρακαλώ όλους να περιορίσουν το χρόνο ομιλίας τους. Καταλαβαίνετε τους χρονικούς περιορισμούς που έχουμε. Σας δίνω το λόγο, κυρία Άννα Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της κυρίας Γιανακουδάκη μιλάω και γι' αυτό μιλάω και αγγλικά. Ευχαριστεί την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότησης. Πιστεύει ότι είναι ένα πολύ καλό σημείο κίνηση για το θέμα αυτό και να γνωρίζει ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ για να προσφέρει μια καλή γνωμοδότηση στην ΕΜΚΟ. Όπως η κυρία Γιανακουδάκη είπε και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, τα κύρια σημεία ανησυχία τη είναι το γλωσσικό ζήτημα. Όπω ε, και το θέμα τη προειδοποίηση επίσης. Θεωρεί ότι είναι ζωτική σημασία να συμπεριλάβουμε μια καλύτερη ρύθμιση για την ε, επιτυχή ολοκλήρωση πιλωτικών προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με την ε, υγεία και όπου περιλαμβάνεται το θέμα της επαγγελματικής ταυτότητας. Όπως λένε πολλοί συνάδελφοι, οι υποχρεωτικά πιλωτικά προγράμματα μπορεί να δημιουργήσουν ε, ένα σύστημα διπλών δύο ταχυτήτων. Γιατί θα υπάρχουν εκείνοι που δουλεύουν με επαγγελματική ταυτότητα και εκείνοι που δουλεύουν χωρίς. Είναι Πιο σημαντικό όμως το θέμα της ε, αμέλειας που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους ίδιους τους ασθενείς. Γι' αυτό θα πρέπει από πριν να έχουν διευκρινιστεί όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε τις τομές και τις διαδικασίες που χρειάζονται για να εισαχθεί το σύστημα της επαγγελματική ταυτότητας Εξού και υποβάλλει την τροπολογία της 33. Αυτά από τη να Γιανακουδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ζέμπα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Άνια Βάιτ Κέρμπερ για τη δουλειά της και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι πολίτες της Ευρώπης ακριβώς περιμένουν από εμά να βελτιώσουμε τη διαφάνεια αυτού του συστήματος, να κάνουμε αυτό το σύστημα περισσότερο κατανοητό προς τους πολίτες. Αν θέλουμε να έχουμε κινητικότητα στην Ευρώπη, πρέπει να μπορούν να ε, αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα και βλέπουμε ότι ε, σε μερικές χώρες τα συστήματα τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν, υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρθηκε ως διτό σύστημα παράλληλης ε, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης σε ορισμένες χώρες και θα πρέπει ε, τα διαφορετικά συστήματα να είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ε, συμβαστική τροπολογία 8, δυστυχώ δεν την υποστηρίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες και η εκπαίδευση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να αποκομίσει μόνο στο σχολείο, αλλά και από πολλούς τομείς γενικής παιδείας και βλέποντας και το σύστημα ε, της ε, υγείας ε, στις χώρες που έχουν αυτή τη θεωρητική εκπαίδευση των 10 ετών και πρακτική στη συνέχεια εκπαίδευση 2 ετών, βλέπουμε ότι λειτουργεί το σύστημα αυτό πάρα πολύ καλά. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και τα θέματα της επικουρικότητας για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή λύση στην τροπολογία 8. Ευχαριστώ πολύ. Καρλ Χάιντς Φλόρενς. Μόλις μπαίνει ο κύριος Φλόρενς. Α, δεν θέλει να λάβει το λόγο ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Άνια Βάισκεβο για την δουλειά που έκανε για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να μιλήσω για την συγκεντρωτική τροπολογία 8. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και πολλά ερωτηματικά για το κατά πόσο πρέπει να βάλουμε μια ελάχιστη ηλικία για να μπορεί κανείς ε, να μπει στην ε, ε, εκπαίδευση των νοσηλευτών και στην πρακτική εκπαίδευση και ενασχόληση με τους ασθενείς. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι αν θα πρέπει να έχουμε μια ελάχιστη σχολική εκπαίδευση είναι καλή ε, η έκθεση και πρέπει να διευκρινίσουμε το ερώτημα του αν χρειάζεται και κάποια τροποποίηση της νομοθεσίας των κρατών μελών αν υπάρξει μια τέτοια πρόταση της Επιτροπής. Η απάντηση είναι ότι ναι, πρέπει να τροποποιήσουν τα κράτη-μέλη τις διατάξεις τους. Κράτη-μέλη τα οποία μέχρι τώρα έχουν ένα επιτυχημένο σύστημα παράλληλης ε, θεωρητικής και πρακτικής ε, άσκησης θα πρέπει να αλλάξουν αυτό το επιτυχημένο σύστημα για να προσαρμοστούν στο σύστημα που προτείνει η Επιτροπή και το ερώτημα θα πρέπει να είναι όχι ποια είναι η εκπαίδευση, αλλά τι την κάνουμε μετά αυτή την εκπαίδευση. Το αποφασιστικό σημείο, το καθοριστικό σημείο είναι το τι μαθαίνει κανείς. Ε, και εγώ ως γιατρός ε, διδάχθηκα ότι η εκπαίδευση των νοσηλευτών μερικές φορές άξιζε περισσότερο από τη δική μου ακαδημαϊκή εκπαίδευση και γι' αυτό είμαι υπέρ αυτής της τροπολογίας. Ευχαριστώ πολύ έχουμε Ροτ Θα μιλήσω αγγλικά για να απευθυνθώ και στην Αντωνία Παρβανόβα. Η συγκεντρωτική τροπολογία 8 για μένα είναι καθοριστική σημασία και πιστεύω ότι είναι εντελώ ασφαλμένη η προσέγγιση του να θεωρείται ότι μια νοσοκόμα θα πρέπει, ένα νοσηλευτή θα πρέπει να κάνει, ε, να πάρει πτυχίο bachelor's ή master's. Είναι εντελώ ασφαλμένη αυτή η άποψη. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να γίνει κανεί γιατρό. Θα είχαμε μόνο γιατρού, δεν θα είχαμε νοσηλευτέ. Θέλουμε να έχουμε νοσηλευτέ που να είναι σε θέση και να είναι και πρόθυμοι να διεκπαιρεώσουν τα συνήθη καθήκοντα που απαιτούνται από του νοσηλευτέ σε ένα νοσοκομείο. Πιστεύω ότι είναι σφαλμένη η δική σα προσέγγιση και είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αυτό το, έχει δίκιο ο Πέτερ Λίζε. Αυτά τα οποία μαθαίνει κανείς στην εκπαίδευσή του μετά το σχολείο, μετά τη σχολική εκπαίδευση, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Και θα πρέπει ε, κάποιος να έχει τη βασική σχολική εκπαίδευση μέσω επίπεδου και γι' αυτό είπα ότι πρέπει μετά τα 16 να μπορεί κανείς να κάνει την πρακτική άσκηση. Αυτό ισχύει και στην ε, ε, Γερμανία, να είναι κανείς 16 ετών για να μπορεί να πάει σε μια ειδική σχολή σε ένα φάχοχσούλε, σε πανεπιστημιακού επίπεδου, ανώτερη εκπαίδευση τέλο πάντων για να επιτρέψουμε την κινητικότητα των νοσηλευτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναγνώριση προσόντων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους νοσηλευτές και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την τροπολογία 8. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι το πιο επίμαχο σημείο. Αυτή η συμβαστική τροπολογία αριθμός 8 ακριβώς γιατί έχει να κάνει με τις ε, απαιτήσει που ισχύουν στις διάφορες χώρες μας. Υπάρχουν χώρες όπου υποχρεωτική εκπαίδευση για όλους είναι 12 χρόνια. Είτε θέλει κανείς να γίνει νοσοκόμος, είτε θέλει να γίνει μηχανολόγος, είτε θέλει να γίνει επιχειρηματίας ή ε, μηχανικός σε συνεργείο. Αλλά αυτό το 12 χρόνια δεν ε, σχετίζεται απόλυτα με το επάγγελμα αυτό που απαιτεί τεράστια υπευθυνότητα και που είναι του νοσηλευτή. Τα 12 χρόνια γενικής εκπαίδευσης ε, λοιπόν έχει να κάνει με αυτό. Και είναι αλήθεια ότι η επαγγελματική εμπειρία είναι σημαντική και ότι ένα ειδικό σχολείο είναι απαραίτητο. Αλλά αυτό ισχύει για όλες τις, όλα τα επαγγέλματα και όχι μόνο για τους ειδικούς για την ε, πληροφορική. Κάθε φορά υπάρχουν ε, δεξιότητες οι οποίες πρέπει να ε, αποκτηθούν μέσω της ειδική κατάρτισης. Εγώ προτείνω να παραμείνουν τα 12 χρόνια. Ευχαριστώ. Ο Κρυς Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Εγώ παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση και είμαι λίγο εκτός, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή η νοσοκόμοι θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, ε, συγκεκριμένη κατάρτιση. Ε, στη χώρα μου φαίνεται να αναπτύσσεται ένα είδος, ε, μάλλον οι νοσοκόμοι, να είναι στην ουσία εκπαιδευόμενοι γιατροί και να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ε, πολλοί θεωρούν ότι είναι νοσοκομιακή εργασία, ενώ στην ουσία είναι βασική ε, συνοδεία, θα το έλεγα εγώ. Εγώ πιστεύω πως οι νοσοκόμοι πρέπει να έχουν ειδικέ δεξιότητες και βέβαια γνώσεις βασικές, βασικής εκπαίδευσης και να κερδίζουν μετά δεξιότητες και προσόντα μέσω της δουλειάς τους στα, στα νοσοκομεία. Δηλαδή, τι νόημα έχει να έχεις ε, πτυχίο γεωλογίας αν μετά πας να γίνεις ζωκόμος. Ευχαριστώ πολύ και θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια την Άνια Βάις Κέρμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Πάλι για την συγκεντρωτική συμβαστική τροπολογία θέλω να μιλήσω. Η κυρία Παρβανόβα είπε ότι οι περισσότερε επαγγελματικές ομάδες και επαγγελματικοί σύνδεσμοι είναι υπέρ των 12 ετών. Και εδώ θα πρέπει να πω ξεκάθαρα για τη Γερμανία ότι το συνδικάτο Verdi που εκπροσωπεί τους περισσότερους νοσηλευτές ξεκάθαρα μίλησε κατά της ε, επιμήκυνσης στα 12 έτη. Γιατί αυτό θα απέριπτε πολλούς νέους που θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα μετά τα 10 έτη. Η συμβαστική τροπολογία στο 8 δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα για αυτούς που έχουν περισσότερα από 10 χρόνια εκπαίδευσης. Μπορούν να διατηρήσουν το σύστημά τους. αυτοί οι οποίοι έχουν ένα είδος εκπαίδευσης ε, το οποίο λειτουργεί μπορούν να παραμείνουν σε αυτό το σύστημα. Επιμένω και γι' αυτό εκφράζομαι με τόσο πάθος υπέρ της τροπολογίας 8. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη συμβαστική λύση και θα δώσουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την ΙΜΚΟ γιατί πιστεύω ότι αυτή την πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ την Άνια Βάις Αύριο θα το ψηφίσουμε. Μας πιέζει ο χρόνος όμως και πρέπει να περάσουμε στην έκθεση Westlund. Και ελπίζω αύριο να πάνε όλα καλά αύριο, Άνια. όσον αφορά την τροποποίηση αυτής της οδηγίας. Λοιπόν, Ευχαριστώ πολύ και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα δώσω το λόγο στην Όσα Βέσλολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, περιμένουμε ο κόσμος να γνωρίζει τι τρώει. Θα έπρεπε να γνωρίζει επίσης τι περιέχουν ε, τα καλλιντικά τα οποία χρησιμοποιεί ή τι υπάρχει μέσα στα έπιπλα που έχουν στο σπίτι τους. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κάποιος έχει πάρει την ευθύνη και έχει φροντίσει ώστε να μην εκτίθενται σε χημικές ουσίες. Και ποιοι είναι αυτοί, εμείς είμαστε αυτοί. Είναι πολύ βασικό προκειμένου να λειτουργεί επίσης και η εσωτερική αγορά. Η Γαλλία, η Δανία έχουν επιλέξει και έχουν υιοθετήσει εθνική νομοθεσία όσον αφορά τι ορμόνε, για παράδειγμα. Ακριβώς γιατί δεν το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό μέσα στη δικιά μου την έκθεση είναι το ότι σήμερα γνωρίζουμε αρκετά πράγματα προκειμένου να δράσουμε και να αντιμετωπίσουμε τους ενδοκρινικούς διαταρακτές. Γνωρίζουμε δηλαδή αρκετά πράγματα για να μπορέσουμε σιγά σιγά να τους απαλείψουμε. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι τέτοιοι ενδοκρινικοί διαταράκτες μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό που δημιουργούν προβλήματα στην αναπαραγωγή, ε, μειώνεται δηλαδή δυνατότητα αναπαραγωγής ή αυξάνονται οι περιπτώσεις διαβήτη. Οι γυναίκες επίσης που υποφέρουν από καρκίνο του μαστού διπλασιάστηκε από το 1980 στον Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που εξηγούν την εξέλιξη αυτή. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν ε, πολλοί λόγοι. Η διατροφή, το στρες, η έλλειψη άσκησης κλπ. κλπ. Είναι πάντως γεγονός, έχει αποδειχτεί δηλαδή από την επιστήμη, ότι οι ενδοκρινικοί ε, διαταρακτές και τα χημικά προϊόντα παίζουν κάποιο ρόλο στις εξελίξεις αυτές. Πόσο σημαντικό είναι αυτό ο ρόλο. Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα σε μια συγκεκριμένη ουσία και μια ασθένεια. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Γιατί η ασθένεια εμφανίζεται μερικές φορές πολύ αργότερα μετά την έκθεση του ατόμου στην χημική ουσία. Έπειτα ακόμα και το έμβριο ε, εκτίθεται σε τέτοιους παράγοντες και δεν εκτίθεται με τον ίδιο τρόπο την έκτη εβδομάδα κύσης όπως και την 16η. Οι ενδοκρινικοί διαταρακτές δρούν μάλιστα ακόμα και σε πολύ χαμηλές δόσεις και μερικές φορές είναι πιο βλαβεροί σε χαμηλή δόση, σε μικρή δόση. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν ε, ομάδες ιδιαίτερα ευάλωτες αυτούς. Οι γυναίκες μάλιστα σε ηλικία αναπαραγωγή είναι πολύ σημαντικές για την αναπαραγωγή, γι' αυτό και πρέπει να τις προστατεύσουμε όλου ιδιαίτερω. Είναι αλήθεια επίσης ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις οικοδομές είναι ε, ουσίες στις οποίες εκτίθεται όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και πρέπει να ρυθμίζονται πολύ αυστηρά. Πρέπει να βασιζόμαστε στην αρχή της πρόληψης. Το ότι δεν γνωρίζουμε δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν κοινά κριτήρια που να καθορίζουν ποιοι είναι αυτοί οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και να γίνουν δοκιμές ώστε να ξέρουμε ποια είναι, ποιες είναι αυτές οι χημικές ουσίες που μπορεί να αποτελέσουν ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ποιε είναι ουσίες αυτές δηλαδή που μπορεί να κρυθούν επικίνδυνε και που γι' αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να παληθούν. Ο εισαγωγέας πρέπει να αποδεικνύει ότι η ουσία που εισάγει είναι ασφαλή και όχι οι κρατικές αρχέ. Δεν πρέπει εκείνες να αποδείξουν ότι είναι επικίνδυνη ουσία όπως ισχύει σήμερα. Πρέπει επίσης να περιορίσουμε την έκθεση κυρίως των νέων σε τέτοιου είδους ουσίες και να ενισχύσουμε άρα τους κανόνες ε, στα τρόφιμα. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν και αυστηροί κανόνες για τα εφάσματα. Τα εφάσματα ακουμπούν στο δέρμα μας. Όπως επίσης να προσέξουμε, όπως σας είπα και πριν, και τα οικοδομικά υλικά, γιατί είναι υλικά τα οποία παραμένουν και ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι στα αγγλικά, στην παράγραφο 4, υπάρχει ένα λάθος. Πρέπει να λέει hazard assessment και όχι risk assessment. Hazard αντί για risk. Αυτά. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ την Εμίλια Ρωμάνο αλλά και την Έλια Ρώμακ την βοηθό μου και από εδώ και πέρα περιμένω τους σκιώδεις εισηγητέ αλλά και τους υπόλοιπους που βρίσκονται στην αίθουσα για να μου πούνε πώς πιστεύουν ότι μπορεί να βελτιωθεί παρατέρω η εκθέση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Κρίστα Κλάση έχει το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ την Οσοβέ Λούντι για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία νομίζω ότι έχει σχέση και με τη συζήτηση που κάναμε για την ποιότητα των υδάτων. Βλέπουμε ότι συνεχώς υπάρχουν νέες ουσίες, ε, τις οποίες ε, παρατηρούμε, οι οποίες εισάγονται. Βλέπουμε ότι προκαλούν κάποιες τροποποιήσεις είτε στον άνθρωπο είτε στη φύση και αυτό θέτει διάφορα ερωτήματα υπάρχει ένα παλιό απόφθεγμα μεταξύ των αγροτών που λένε ότι ό,τι δεν ξέρουν οι αγρότες δεν υπάρχει. Ε, αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα οποία έχουμε κάνει, δεν θα φτάναμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του ε, τι κινδύνους ενέχει η καινοτομία οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ε, είναι ουσίες που πρέπει να λυθούν ε, ιδιαίτερα σοβαρά γιατί υπάρχουν και σε προϊόντα φυτοπροστασίας ε, και σε διάφορα φυτά όπου δρούν ως ορμόνες όπως τη σόγια ή στον καφέ και είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η κατάσταση. Πολύ σωστά περιγράφει η κυρία Βέσμου στην έκθεσή της ότι υπάρχουν ε, διάφορες ε, συνέπειες όπως είναι ε, η χειρότερη κατάσταση του σπέρματος παραδείγματος χάρη, οι διάφορες παραμορφώσεις. Θα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα κριτήριο με ένα συγκεκριμένο όριο, ένα κατόφλι το οποίο οποίο θα θέσουμε και θα πρέπει να ισχύει, ένα cut-off ε, όριο. Ε, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και γι' αυτό θα θέλαμε επιστημονικές συμβουλές ε, και αυτό ζητούμε από τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Η επιστήμη προχωρεί όλο και περισσότερο, αλλά δεν μπορούμε πάντοτε να βρούμε τις ε, ε, επακριβείς ποσότητες ε, διήθησης στο έδαφος, παραδείγματος χάρη. Στο σημείο 5 όμως έχουμε ένα παράδειγμα, ένα σημείο στο οποίο δεν είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο θεσπίζουμε για τα κριτήρια. Θέλουμε θα θέλαμε να μπορούμε να προσδιορίσουμε το τι είναι ένας ανεπηρέαστος οργανισμός, αλλά ε, οι άνθρωποι και τα φυτά και τα ζώα είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο και δεν μπορούμε να πούμε τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι φυσιολογικό και αυτό να το ορίσουμε με ένα συγκεκριμένο ορισμό θέλουμε μια διαδικασία αξιολόγησης ε, που να θεωρείται πολιτικά αποδεκτή ε, και ένας διεθνής ορισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το τι σημαίνει ε, επιπτώσεις και επικινδυνότητα σε ένα πραγματικό οργανισμό και όχι μόνο in vitro. Τα φάρμακα ε, δρούν επί των ε, ορμονών ε, και ορισμένα φάρμακα είναι πιο ισχυρά από άλλα και γι' αυτό χρειαζόμαστε διαφορετικές κατηγορίες για την δραστικότητα και για την επικινδυνότητα. Θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τους ορμονικούς διαταράκτες και πολύ συχνά οι επιπτώσεις τις οποίες υποστηρίζει ένα εργαστήριο δεν υποστηρίζονται από ένα άλλο εργαστήριο. Υπάρχουν δηλαδή αντιφατικά αποτελέσματα. Πολύ συχνά δεν έχουμε αντικειμενικά στοιχεία, αντικειμενικές τιμές τις οποίες μπορούμε να βασιστούμε. Πρέπει λοιπόν και οι μέθοδοι αξιολόγηση ε, να οριστούν πολύ προσεκτικά. Ευχαριστούμε, Κρίστα Κλά, η κυρία Λεπάζ, αλλά μισό λεπτό παρακαλώ, περιμένετε. Ε, γιατί έχουμε τη σκιώδη εισηγήτρια και τους υπόλοιπου ομιλητέ και μετά θα κλείσει ο κατάλογο των ομιλητών, αν δεν προσταθεί κάποιο. Haben wir alle. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Βέστλοντε για το εξαίρετο έργο της που προχωρά προς πολύ σωστή κατεύθυνση αλλά που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ενισχυθεί σε πολλά σημεία. Καταρχήν Χαίρομαι που βλέπω ότι η αρχή της προφύλαξης εδώ αναφέρεται και μάλιστα υπενθυμίζεται και Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε στο τι είναι η αρχή της προφύλαξης και όχι στις ε, διάφορες ερμηνείες που κάποιες φορές έχουν και χαρακτήρα καρικατούρας. Ε, είναι στοιχεία πολλές φορές όπου πολλές φορές μιλάμε για αρχή προφύλαξης αλλά στην ουσία πρόκειται για απλή πρόληψη. Από τη στιγμή λοιπόν που χρειάζεται να διερωτηθούμε Εντάξει, αλλά να ζητήσουμε ε, παληθευμένα στοιχεία νομίζω πως δεν είναι ένα τέτοιο, δεν έχει νόημα. Η αρχή της προφύλαξης σημαίνει αρχή έρευνας για να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μπορεί και σε απορίες μπορεί να έχουμε. Τώρα, στο τι υπάρχει διαθέσιμο, το γεγονός ότι ανατρέχουμε στις, σύγχρονε στις σύγχρονες και πρόσφατες έρευνες είναι καλή ιδέα και ότι αυτό το στοιχείο θα πρέπει να ενισχυθεί. Να υπογραμμίσω δε εδώ ότι στη Γαλλία η υγειονομική μας υπηρεσία αναγνώρισε την ανάγκη παρέμβασης για διάφορα στοιχεία όπως το, την δυσφενόλη και εκεί για να το καταφέρει αυτό έλαβε υπόψη όλες τις μελέτες που υπήρχαν επιτάπητες συμπεριλαμβανομένων αυτών των οποίων τα πειραματικά πρωτόκολλα δεν αντιστοιχούσαν αναγκαστικά πάντοτε στις σωστές πρακτικές, ορθές πρακτικές των εργαστηρίων. Και πολλοί εμπειρογνώμονες θεωρούν σήμερα πως τα τυποποιημένα τεστ έχουν ξεπεραστεί γιατί είναι δυνατόν να μην ανοιχνεύσουν ε, την επιρροή στοιχείων και ουσιών όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Ε, τώρα, η προσέγγιση της εισηγήτριας για τις ουσίες που δεν έχουν κατώτατο όριο θα πρέπει να ορίσουμε τις τιμές αυτές και θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη τις συνδυασμένες επιπτώσεις, επιπτώσεις των κοκτέιλ, ε, ένα θέμα για το οποίο συχνά μιλάμε εδώ, αλλά που είναι πραγματικό ζήτημα. Τέλο, η συγγήτρια καλεί την Κομισιό να υποβάλει την ε, νομοθεσία σε συστηματική εξέταση και σε περίπτωση που αυτό χρειάζεται να υποβάλει νέα νομολογία ώστε να μειωθεί η έκθεση στον πληθυσμό. Υποστηρίζω απόλυτα αυτό το διάβημα. Σα ευχαριστώ. Μισελ Μπεζή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια για την έκθεση αυτή, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και για αυτές τις προτάσεις. Εγώ είχα ένα ερώτημα, μια διευκρίνηση από πλευρά της Κομισιόν θα επιθυμούσα, διότι εδώ και ένα χρόνο υπό την αιγίδα της ΓΔ περιβάλλον ε, ζητήθηκε να αποσαφενιστεί η στρατηγική και οι επιστημονικές και οι πολιτικές επιπτώσεις σε σχέση με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και μαθαίνουμε πως η Κομισιόν ζήτησε την έκθεση, μια άλλη έκθεση στην ΕΦΣΑ. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος επικάλυψης ανάμεσα σε όλο το πλωστάσιο που ήδη έχει γίνει από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ περιβάλλον που, συνεδρια... που συνδυάζεται η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ υγεία, η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Χημικά Προϊόντα, οι διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων που ένα σωρό συνεδριάσεις και η Κομισιόν τώρα ξαναζητά από την ΕΦΣΑ να ξανακάνει την ίδια μελέτη. Δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών, γιατί ζήτησε τέτοια μελέτη η Κομισιόν στην ΕΦΣΑ. Δεύτερον, η ΕΦΣΑ ξέρετε ότι υπήρξαν διάφορες συγκρούσεις συμφερόντων εκεί, γιατί δεν υπερψηφίστηκε η απαλλαγή της εδώ και λίγο έγινε αυτό, για να διευκρινιστούν οι σχέσεις της με τη βιομηχανία. Οπότε, το διακύβευμα εδώ είναι να έχουμε ένα πολύ καλό ορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Και σε σχέση με τα όσα λέγατε, κυρία Κλάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό είτε είναι η γαμαδέλτα περιβάλλον, είτε είναι οι περιγνώμονε των κρατών κτλ. να κάνουν όσο γίνεται ευρύτερο ορισμό. Γιατί, Γιατί οι ενδοκρινικοί διαταράκτε δεν έχουν τι ίδιε επιπτώσει όπω άλλα μόρια. Δεν είναι η δόση που φτιάχνει το δηλητήριο εδώ. Περισσότερο είμαστε σε έναν γραμμικό τομέα. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι σε πολύ μικρές δόσεις μπορεί ακριβώς να υπάρξουν διαταραχέ στο, στο μεταβολισμό και εδώ, και εδώ έρχομαστε όσα έλεγε η Κορίν Λεπάζ, δεν είμαστε τόσο στο θέμα της προφύλαξης όσο στο θέμα της πρόληψης. Δηλαδή υπάρχουν πάνω από 700 μελέτες που έχουν δείξει τη σύνδεση ανάμεσα σε γενετικές ε, ε, και ε, σχηματισμούς και διάφορες άλλες διαταραχές σε πολύ μικρές δόσεις, πολύ μικρές δόσει. Και έπειτα έχουμε και τις ε, παρενέργειες των διαφόρων κοκτέιλ. Είμαστε σε άλλη υπόθεση, δηλαδή επιστημονική. Και θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε τα προϊόντα τα οποία φτιάχνουν οι βιομήχανοι είναι ενδοκρινική διαταράκτηση ή όχι. Είναι επίγον, είναι επίγον γιατί είναι επίγον απέναντι στα παιδιά αλλά και στι εγγύου γυναίκε. Η Γαλλία και η Δανία ήταν πολύ δραστήριε. έφτιαξαν μια νομοθεσία για να εμποδίσουν α πούμε από τα 0 μέχρι τα 3 έτη τη δυσφενόλη, αλλά πρέπει περισσότερο να προχωρήσουμε αν δεν θέλουμε να ε, παίρνουν τέτοιου ενδοκρινικού διαταράκτες οι έγκυε γυναίκε Και να ζητήσω λοιπόν από την Κομισιόν σε θα, πώ θα, πώς θα ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία η έκθεση που ζητήσατε. Και από διεθνή άποψη όλοι αναγνωρίζουν ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτε έχουν επιρροή. Είτε βάζουμε λεφτά στην υγεία λοιπόν Είτε ε, ε, με ένα σωστό ορισμό υποχρεώνουμε τους βιομήχανους, τους φάρμακοβιομήχανους, εφόσον φτιάχνουν τέτοια προϊόντα, να εξακριβώνουν αν ναι ή όχι εμπίπτουν στους ενδοκρινικούς διαταράχτες και αν ναι να τα απαγορεύουν. Ευχαριστώ η κυρία Σόζα. Όχι. Αφού δεν θέλετε το λόγο, Άννα δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του Προέδρου μας που δεν είναι παρόν και γι' αυτό εγώ θα σας παρουσιάσω τη θέση της ομάδας μας. Εκτιμούμε ότι η έκθεση αυτή δεν είναι αρκετά ισορροπημένη και δεν έχει βασιστεί στις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Θα πρέπει να ε, συμφωνήσουμε για τον ορισμό ενός, του τι είναι ο ενδοκρινικός διαταράκτης. Ε, πρέπει να αναφερθούμε στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που ορίζει αυτούς τους διαταράκτες ως ουσίες που έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Η έκθεση σχετική λέει ακριβώς πως αυτό το είδος ε, γνώσεων δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν αρκετές γνώσεις και τα συμπεράσματα βγαίνουν επί τη βάση ατελών γνώσεων. Εμείς λοιπόν ανησυχούμε για το Ε, μάλλον αμφισβητούμε ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις μέχρι ότου αυτό αποδειχθεί με στέρες επιστημονικές βάσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να έχουμε μια προσέγγιση που βασίζεται σε αποδείξεις. Ελπίζουμε λοιπόν πως η έκθεση αυτή θα τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ, Άννα Ρόσμπα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ την εισηγήτριά μας για την εξαιρετική της έκθεση, η οποία είναι σαφέστατη και που ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να ενεργήσουμε εδώ και τώρα. Να θέσουμε απαιτήσει. Η παρέμβαση δε της κυρίας Ρόσμπακ ήταν κάπως παράξενη. Διότι δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι η εδοκρινική διαταράκτηση είναι επικίνδυνη. Αυτό το οποίο είναι δύσκολο να καθοριστεί είναι ποια είναι τα όρια από τα οποία και πέρα γίνονται αισθητές οι αρνητικές παρενέργειες. Και γι' αυτό και θεωρώ, κυρία Westlund, ότι η έκθεσή σας είναι εξαιρετική. Μπορούμε ωστόσο να την ενισχύσουμε παρουσιάζοντας ένα χρονοδιάγραμμα στην Κομισιόν για την επεξεργασία της στρατηγικής και για την ανάληψη δράσης. Και έπειτα θα πρέπει να δούμε μήπως ήταν ενδιαφέρον να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό κέντρο που θα είναι αφιερωμένο στους δοκρινικούς διαταράκτες. Υπάρχει τέτοιο κέντρο στη Δανία και νομίζω ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουμε ε, αυτή την εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της γνώσης ε, επί του θέματος αυτού. Τούτου λεχθέντος είναι πραγματικά εξαιρετική έκθεση και ελπίζω πως δεν θα αποδυναμωθεί. Ο κύριος Σλούτερ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ρόζα για αυτή την εξαιρετική έκθεση και να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονό, στην συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο σχετικά. Μιλάμε τώρα για τις διάφορες κατηγορίες χημικών προϊόντων, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι το κατά πόσο το προϊόν είναι, να αποφασιστεί κατά πόσο είναι επικίνδυνο το προϊόν και έπειτα να δούμε σε ποιες σε ποσότητες καθίσταται πιο επικίνδυνο. Τώρα, όσον αφορά του ορισμούς. δεν υπάρχει κάποια τέλειος ορισμός για όλους αυτούς τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν οι ορισμοί, λαμβάνοντα υπόψη τις άλλε οδηγίες που διέπουν αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια πως η συζήτηση είναι περίπλοκη, είναι δηλαδή σημαντικό να μην μετατραπούν όλα αυτά ε, σε μια απλή έκθεση πρωτοβουλία. Θα πρέπει να ενεργήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προστατευτεί ο καταναλωτή. Προσπαθεί κανεί να φάει υγιεινά, τρώει μια σαλάτα με ντομάτα και αγκούρι και πρασινάδες όμως αυτά είναι τα τρία λαχανικά όπου ε, βρίσκει κανείς την πιο μεγάλη συγκέντρωση ενδοκρινικών διαταρακτών. Όλος ο κόσμος όμως θεωρεί ότι είναι υγιεινή η σαλάτα. <laughs> μπορεί κανεί να αγοράζει βιολογικά προϊόντα, εντάξει, αλλά πολύ πιο ακριβά. Είναι δύσκολο ωστόσο να βρει κανεί χωρί δυσφενόλη τέτοιου είδους ε, σαγητά. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή διαδικασία. Έγινε και μία ακρόαση, νομίζω, ε, που από ό,τι άκουσα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν οι εμπειρογνώμονες παρόντες που έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα υπό έλεγχο και υπήρχαν και οι άλλοι που έθεταν ε, τα ανοιχτά ερωτήματα που έλεγαν ότι οπωσδήποτε χρειάζεται να προχωρήσουμε και στην έρευνα και στις ρυθμιστικές διατάξεις. Νομίζω ότι η έκθεση δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνει η Επιτροπή. Θέλουμε έναν ορισμό το άρθρο 3 τίθεται το ερώτημα του αν θέλουμε μια ταξινόμηση, όχι μόνο έναν ορισμό, αλλά και μια ταξινόμηση ανάλογα με ε, το μέγεθος της επιβάρυνσης. Μετά στο άρθρο 4 ε, ζητάμε μια αξιολόγηση κινδύνου εδώ θα συμφωνούσα με όσους λένε ότι υπάρχει η αρχή της προφύλαξης και θα πρέπει να είναι συνολική η αξιολόγηση κινδύνου, όχι μόνο δηλαδή στα σημεία όπου υπάρχουν σαφείς ε, ενδείξεις επιδείνωσης, αλλά με την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Μετά στο άρθρο 5 αναφέρεται ο κανονισμός REACH, ε, και αναφέρεται και η υποκατάσταση, το substitution που πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του REACH όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Είναι καλή αυτή η έκθεση και νομίζω με βάση αυτήν την έκθεση μπορούμε να δουλέψουμε περαιτέρω και η Επιτροπή θα πρέπει να μας πει πώς θα χειριστεί τα θέματα αυτά από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής ο επικεφαλής ε, της ε, μονάδας, ο κύριος Χάνσεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω δύο λόγια για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και θα προσπαθήσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας για το έργο της ΕΦΣΑ. Αναθερούμε την τρέχουσα στρατηγική πρόθεσή μας είναι να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση αυτή κατά τη διάρκεια του 2012, ακόμα το πολύ στις αρχές του 2013, ώστε να προχωρήσουμε μετά την επιτυχία της προηγούμενης στρατηγικής. Συνεχίζουμε λοιπόν βάσει της στρατηγικής ε, αυτής και στόχος μας είναι ο Μάρτιος ή ο Απρίλιος της επόμενης χρονιάς προκειμένου να έχουμε μια νέα στρατηγική που θα βασίζεται βέβαια στις εμπειρίες μας από την προηγούμενη. Συγχρόνως σκοπεύουμε να έχουμε έτοιμη και μια πρόταση για τον ορισμό και τα κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες στα μέση της χρονιάς, δηλαδή του χρόνου, μετά το Μάρτιο-Απρίλιο, θα την έχουμε και αυτή την πρόταση. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν Δουλέψαμε πολύ σε ομάδες τα δύο τελευταία χρόνια με επιστήμονες από όλες τις πλευρές. Η δουλειά αυτή για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες γίνεται συγχρόνως με διαβούλευση με το κοινό που αποκορύφθηκε με μία διάσκεψη στα μέσα του 2012 η οποία κατέληξε λίγο πολύ στην ίδια γραμμή με αυτή που βλέπουμε και στα εισαγωγικά σημεία της ε, έκθεσης της κυρίας Βέσλαν. Το συμπέρασμα δηλαδή ήταν ότι έχουμε συλλέξει πολλή γνώση και πολλά επιστημονικά δεδομένα μέχρι τώρα και ότι βλέπουμε πως από τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η χρησιμοποίηση των επιστημονικών αυτών δεδομένων. Για να έρθω τώρα στις αποσαφηνίσεις όσον αφορά τη δουλειά της ΕΦΣΑ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το διευκρινίσω αυτό. Γιατί θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί όντω ότι πρόκειται για επικάλυψη προσπαθειών. Δεν είναι όμως αυτή η πρόθεσή μας και ούτε ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς ακολουθούμε τη διαδικασία που σας εξήγησα. Αυτό είναι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΗ, αλλά συνεργαζόμαστε συγχρόνως στενά με τις άλλες γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με χημικές ουσίες. Ζήτησε τώρα η Επιτροπή την άποψη της ΕΦΣΑ για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες στα πλαίσια της εντολής της ΕΦΣΑ. έχει νομική, υπάρχει νομική υποχρέωση των συναδέρφων από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ να ζητούν την γνώμη της ΕΦΣΑ όταν προετοιμάζουν κάποια θέματα. Και αυτό ακριβώς συνέβη και με την ΣΑΝΚΟ και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες στα πλαίσια της νομοθεσίας που ετοίμαζε για τα παρασιτοκτόνα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ζητούμε τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Δεν πρόκειται όμως για ε, καμία επικάλυψη. Είναι η συνήθις διαδικασία προκειμένου να προχωρήσει η νομοθετική δουλειά για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάντσεν και θα δώσω το λόγο στην εισηγητή, την κυρία Σεβέσλουν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε σε βάθος. Δύο λεπτά από ό,τι βλέπω έχουμε στη διάθεσή μας. Πάντως τέτοιες συζητήσεις θα τις έχουμε και στο μέλλον. Κατά τη γνώμη μου είναι αναγκαίο να παρακολουθούμε από κοντά την επιστημονική έρευνα. Όταν ρωτάμε ερευνητές που ασχολούνται με ενδοκρινικούς διαταράκτες μας λένε φοβερά πράγματα. Υπάρχουν και δύο αναφορές στην έκθεση που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που μιλάει για την κατάσταση της έρευνας, για κριτήρια κτλ. Εμείς δεν πιστεύω ότι πρέπει τόσο ρητά να τα αναφέρουμε αυτά, αλλά πρέπει να δίνουμε κάποια ένδειξη. Βλέπετε Πάντως ο επιστημονικός κόσμος πώς ε, βλέπει τα πράγματα. Είναι αλήθεια, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αλλαγές στην υγεία των ανθρώπων, εξελίξεις. Ε, δεν είναι καινούριο αυτό, το συζητάμε εδώ και δεκαετίες. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν έχει ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα. εκτός από το Μπεν Πες, τα μπουκάλια. Κατά τα δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ επήγει το θέμα. Αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι, πρέπει να προχωρήσουμε σε δράση. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία προοδεύει, προχωράει όταν μπορούμε να αντικαθιστούμε επικίνδυνα προϊόντα από άλλα προϊόντα τα οποία προστατεύουν και το περιβάλλον και την υγεία μας. Συνεπώς δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην κοινωνική πρόοδο και την απαγόρευση επικίνδυνων ουσιών. Αντίθετα αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 16 Νοεμβρίου και στις 18 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κατά πάσα πιθανότητα στην Ολομέλεια η ψηφοφορία θα γίνει τον Απρίλιο του 2013. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συζήτηση και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10 για την ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Σνέλχαρτ την ψηφοφορία.